Um, although uh, <laughs> not all shadows δεν βλέπω να έχουν έλθει όλοι οι σκιώδεις αλλά είναι πάρα πολύ φορτωμένοι με τη σχεδιάταξη γι' αυτό προτείνω να ξεκινήσουμε έχουμε 45 λεπτά για, μια, για ένα γύρο έρωτα απαντήσεων η συμπρόεδρη της Ελληνικής Ομάδας Εμπειρογνωμών για την προστασία των δεδομένων, η ευρωπαϊκή πλευρά ε, θα μας ενημερώσει για το πώς έχει κατάσταση των συζητήσεων με τις Αμερικανικές Αρχές. Συναντήθηκαν όπως γνωρίζουμε τον Ιούλιο δύο φορές και την προηγούμενη εβδομάδα 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην Ουάσιγκτον. Ο κ. Πονέμιτς ε, θα μιλήσει εξ ονόματος Τη αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε την ομάδα εργασίας. Εν συνεχεία θα μπορούν οι συγητές και οι σκιώδες να κάνουν τις ερωτήσεις τους. Θα σας ζητήσω να απαντήσετε και αν έχει μείνει χρόνος. Θα μπορέσουν και άλλοι συνάδελφοι να σας ε, κάνουν ερωτήσεις. Κύριε Νέμιτς, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεδρία της ομάδας εργασία. Ε, είπατε ότι εμεί για την πρώτη συνεδρία, σε αυτή μια διερευνητική συνεδρία για το κατά πόσον θα ήταν σκόπο να γίνονται ή να μην γίνονται τέτοιε συναντήσει. Στη δεύτερη ε, συνάντηση επικεντρωθήκαμε ε, σε ένα αίτημα τη Αμερικανική Πρόεδρο που ήταν ο έλεγχο, η αποπτία και τι μηχανισμοί μπορούν να εγγυηθούν ότι οι μυστικές υπηρεσίε ε, και ε, θα δρούν σύμφωνα με το δίκαιο των Ε, Έχουμε δύο συστήματα, εκτελεστικό έλεγχο, εκτελεστική εποπτεία από τη μία πλευρά και ακούσαμε μία παρουσίαση ε, από το γραφείο Privacy Office ε, των, ε, της αντίστοιχης υπηρεσίας των ΙΠΑ και από την αρχή την εποπτική και όλους αυτούς που ασχολούνται με με το θέμα αυτό και είχαμε και το, την εποπτεία, την κοινοβουλευτική κατά κάποιο τρόπο, από το Κογκρέσο δηλαδή. Υπάρχει ειδική επιτροπή και στη Γερουσία και στο Κογκρέσο. Και μπαίνει και μια άλλη αρχή, τη δικαστική εποπτεία, την είναι αυτή την πρώτη, είναι το Υπουργείο Δικαιοσύνη. Επίση, η Αμερικανική κυβέρνηση επέτρεψε να συναντηθούμε και με τους δύο προέδρους των επιτροπών που έχουν επιφορτηθεί από τον πρόεδρο Ομπάμα ε, με τη διατύπωση προτάσεων για μεταρρυθμίσεις των νόμων ε, περί επιτήρησης και των σχετικών πρακτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας από τους φορείς αυτούς ε, λέγεται P-Club, με τους οποίους συναντηθήκαμε τον πρόεδρό του συγκεκριμένα, ένας φορέας ο οποίος θα πρέπει να επιβλέπει όλες τις αντιδρομοκρατικές δραστηριότητες δε βάση νόμου. Στη ΣΥΠΑ και αναφέρει ε, σε ημερομηνία που προβλέπεται, αλλά δεν θα είναι πάρα πολύ ε, μακριά, πάνω σε τρία θέματα. Πρώτον, αν οι δραστηριότητες ε, των υπηρεσιών της, των ΙΠΑ τηρούν το δίκαιο, αν οι νόμοι με βάση οποίου λειτουργούν είναι συνταγματικοί και τρίτον ακόμη και αν είναι νόμιμες ε, οι συνταγματικέ δραστηριότητε, ή μάλλον και συνταγματικέ, αν αυτέ οι πολιτικέ είναι σωστέ. Και συναντήσαμε επίση, έναν άλλο φορέα που έχει συγκροτηθεί από τον πρόεδρο και ο οποίος θα πρέπει να διατυπώσει προτάσεις για την καλύτερη ε, χρήση της τεχνολογίας και τη συμφιλίωση της εθνικής ασφάλειας ε, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την προστασία των δεδομένων. Ο Πίτερ Σουάιερ είναι ο πρόεδρος. Είναι μια ad hoc που θα αναφέρει εγγράφος γύρω στα τέλη του έτους και προφορικά στον πρόεδρο βέβαια σε δύο εβδομάδες, 22 μέρες από την συνάντησή μας τότε και οι δύο ομάδε μας έδωσαν την εντύπωση ότι έχουν, υπάρχει ένα άνοιγμα, κάποιο άνοιγμα ε, για αλλαγέ. Και το δεύτερο ad hoc σώμα αυτό μα είπαν ότι είναι και μέρο τη εντολή του να εξετάσουν εξωτερική πολιτική, γιατί τόσες ε, υπάρχουν για αυτή. Βέβαια, ζητήσαμε κι εμείς να μας απαντήσουν στις ερωτήσεις μας που είχαν να κάνουν ε, και πάλι με το πεδίο εφαρμογή, ε, με το εύρος και την επίπτωση αυτών των δραστηριοτήτων ε, στους πολίτες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν περιορισμένες. Ουσιαστικά περιορίζονταν στο θέμα της εποπτείας, του, προσπάθησαν να μας καταδείξουν και ήταν και εντυπωσιακό θα ήθελα να σας πω, ότι στο σύστημα των ΙΠΑ υπάρχει πάρα πολύ στενό σύστημα ελέγχων που φροντίζουν σε ένα μεγάλο βαθμό να δρουν με βάση την Αμερικανική νομοθεσία οι υπηρεσίε αυτέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Μωράη, τον εισηγητή, για να σχολιάσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πιο πολλές σκιές παραφώς έχουμε εδώ, πιο πολλούς σκιώδεις εισηγητές δηλαδή, παρά τίποτα άλλο. Θέλω όμως να ευχαριστήσω τον ομιλητή που ήταν σύντομος για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ποια ήταν η ουσία των θεμάτων που συζητήθηκαν στις επαφές αυτές που αναφέρατε και καταρχήν αν υπήρξε η εντύπωση ότι αφορά πάρα πολλούς Ευρωπαίους πολίτες αυτή η δραστηριότητα ή τουλάχιστον οι καταγγελίες αυτές δραστηριοτήτων Έχετε κάποια ιδέα για το οι Ευρωπαίοι πολίτες καλύπτονται από τις διαδικασίες αυτές παρακολούθησης στις ΗΠΑ, μια αίσθηση της σοβαρότητας των πιθανών επιπτώσεων, πόσο, σε τι επίπεδο λεπτομέρειας συλλέγονται πληροφορίες. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ξέρουμε αν αυτό συστήθηκε σε κάποια από τις επαφές σας. Και δεύτερον, μιλήσατε για συστήματα εποπτείας κτλ. Αυτό είναι ενδιαφέρον. Αυτό είναι σημαντικό. Αλλά στην πράξη μπορεί να υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι νόμιμες σε επίπεδο Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά όταν εφαρμόζονται σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάσουν τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματος χάρη η συλλογή δεδομένων μέσα από τα καλώδια οπτικών ινών που φτάνουν στι Ηνωμένες Πολιτείες για το διαδικτυό. Υπήρξε λοιπόν αυτό το ερώτημα σε κάποια από τις συζητήσεις σας που σας απασχόλησε. Δώστε μας περισσότερες λεπτομέρειες αν ήταν τμήμα της συζητήσεως που είχατε. Και επίσης το θέμα του ασφαλούς λιμένα. Αν συζήτησε η ομάδα η Διατλαντική τη δυνατότητα αναθεώρησης των ε, κανόνων για το λεγόμενο ασφαλή λιμένα. Αυτό ήταν μια συμφωνία που έγινε το 2005 και τώρα προφανώς επειδή έχουν αλλάξει τα πρότυπα χρειάζεται ίσως να δούμε κατά πόσον εξακολουθεί να συνάδει με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία το σύστημα αυτό του ασφαλούς λιμένα και ποια είναι και η αντίδραση που υπήρξε για τα θέματα αυτά. Και επίσης αν λάβουμε υπόψη την σημασία των Αμερικανικών εταιριών οι οποίες συνεργάστηκαν με την κυβέρνηση για τα θέματα αυτά. Είδατε οι ΗΠΑ να είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε κάποια αναθεώρηση του ασφαλούς λιμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φως δεν είναι παρόν από το ΕΛΚ. Α, έρχεται, ναι. Θα αφήσουμε τώρα τον κύριο Βος. Και εγώ δεν θα λάβω το λόγο σε σκιώδες, θα μιλήσω στο τέλος. Θα δώσω το λόγο στους πράσινους. Σας ευχαριστώ, λέει ο Γιάνν Άλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και πάλι. Έχω την εντύπωση ότι σε επίπεδο ουσίας τα μέτρα αυτά παρακολούθησης και το ότι κρύπτεται πίσω από αυτά τα μέτρα δεν θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Εγώ Εστιάζω στη δική σας εκτίμηση για το τι έλαβε χώρα στη συνάντηση αυτή. Προς το παρόν είναι φανερό ότι το ερώτημα είναι υπάρχει κάποια πιθανότητα ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι, να αλλάξουμε κάτι και η δική μου εντύπωση είναι ότι ορισμένοι θα πούν ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αλλάξει κάτι γιατί δεν υπάρχει αλλαγή πολιτικής νοοτροπίας στις ΗΠΑ για το θέμα αυτό. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό αληθεύει ή αν πράγματι μπορείτε να διακρίνετε κάποια αλλαγή στην νοοτροπία στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχω δει διάφορες γνώμες για το θέμα. Για τη συμφωνία Φάιζα, το νόμο Φάιζα, ενδεχομένως να υπάρξει μια τροποποίηση στη νομική βάση, γιατί εκεί είναι το πιο σημαντικό για τους Ευρωπαίους. Νομίζω ότι υπάρχει κάποια παρεξήγηση ότι εμείς ως Ευρωπαίοι έχουμε ερωτήματα σε σχέση με την νομιμότητα αυτών των μέτρων παρακολούθησης σε σχέση με την Αμερικανική νομοθεσία αλλά δεν μας απασχολεί καθόλου το θέμα της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Και εδώ χρειάζεται να το διευκρινίσουμε αυτό και θα ήθελα γι' αυτό το λόγο να συζητήσω ποια είναι η κατανόηση, αν υπάρχει κατανόηση, μεταξύ των Αμερικανών για αυτή τη διαφορά που είναι πολύ σημαντική. Ότι ακόμα και αν υπήρξε ένας νόμος <clears throat> για παρακολούθηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί αυτός να παραβιάζει τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου λοιπόν. Ευχαριστώ. Κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που θα πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά αν θέλουμε να παραμείνουμε με αυτή την κατάσταση που τα πράγματα βρίσκονται στο σκοτάδι και είναι ένα μαύρο κουτί ουσιαστικά. Δεν έχουμε λοιπόν βγάλει κάτι σε επίπεδο ουσίας. Σε μένα λοιπόν είναι ουσιαστικό το τι μπορούμε να αποκομίσουμε από τέτοιες επαφές και εξακολουθώ να έχω πάρα πολλές αμφιβολίες για το τι μπορούμε να μάθουμε με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να θέσω κάποια ερωτήματα που εξακολουθούν να έχουν νόημα από τη δική μου πλευρά. Ποιος πα... Πώς γίνεται η παρακολούθηση της εργασίας αυτής της ομάδας, πώς προχωράει αυτή η διαδικασία. Βλέπετε έγγραφα, βλέπετε φακέλους, τι έχετε στη διάθεσή σας. Τι ακριβώς κοιτάτε σε αυτές τις συνεδριάσεις και τι είδους συμπεράσματα μπορείτε να βγάλετε. Με ποιους κανόνες γίνεται η εξέταση των θεμάτων. Βασιζόμαστε στο Αμερικάνικο δίκαιο, στους ευρωπαϊκούς κανόνες, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Και επίσης υπάρχει μια παραδοχή από την πλευρά των Αμερικανών ακόμα και σε ήπιο επίπεδο ότι υπήρξε μια παρακολούθηση. Υπάρχει μια βάση λοιπόν συζήτησης ή είναι κάτι το οποίο δεν το αποδέχονται οι Αμερικανοί. Και στοιχεία θέλω αριθμούς, πολλούς αριθμούς. Ποια είναι τα αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από αυτή τη διαδικασία. Αλλιώς δεν νομίζω ότι έχει νόημα να συζητούμε. Ευχαριστώ και ακριβώς την στιγμή που πρέπει ο κύριος Φως. Κρίμα που δεν μπόρεσα να ακούσω τη δήλωσή σας και σας ζητώ συγγνώμη. Θα με ενδιαφέρε να ξέρω για το ποιες είναι οι εγγύησει που μπορεί να έχει κάποιος από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι δεν γίνεται βιομηχανική κατασκοπή από τη δική τους πλευρά. Και αυτό το λέω γιατί, γιατί η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται από ιδιωτικές εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ γρήγορα, κύριε Κίρκοφ, θέλετε να πείτε κάτι. Όχι τώρα. Θα δώσω το λόγο στη Σόφη Ιντφέλτ. Κύριε Νίμιτς, μην το πάρετε προσωπικά. Αλλά έχω πολύ σκεπτικισμό σε σχέση με την χρησιμότητα αυτού του εγχειρήματο. Δεν νομίζω ότι μιλάμε για ένα απλό διοικητικό θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από μια ομάδα εργασία κρατικών αξιωματούχων, όσο αφοσιωμένο και ικανό να είναι. Και επίση, όπω σχεδόν όλοι οι προηγούμενοι ομιλητέ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώ θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για μια αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πηγαίνει στη Washington για να τους δώσουν μια διάλεξη για το Αμερικανικό Σύνταγμα και την Αμερικανική νομοθεσία. Αυτά μπορούμε να τα διαβάσουμε κι αλλού. Το θέμα είναι να ξέρουμε τι ακριβώ έγινε με εμά, αν έχει παραβιαστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό είναι δική μα ευθύνη και όχι τη Αμερικανική κυβέρνηση. Για την κρίση σα επίση. Είπατε ότι σα κάνανε μια παρουσίαση για του μηχανισμού εποπτεία και εντυπωσιαστήκατε αλλά ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαδικασίας βασίζεται σε μυστικούς νόμους που εφαρμόζονται και ελέγχονται από ένα μυστικό δικαστήριο, ένα δικαστήριο που δεν συνεδριάζει δημόσια. Αν αυτό σας εντυπωσιάζει, τι άλλο σας εντυπωσιάζει και πώς μπορείτε να θεωρήσετε ότι αυτές οι μορφές εποπτείας είναι εντυπωσιακέ, Μου φαίνεται όλη αυτή η ιστορία ότι γίνεται μονάχα για συμβολικούς λόγους δεν θέλει ο κύριο Κίρκοπ να πει κάτι. Θα ζητήσω τον κύριο Νέμιτ να απαντήσει και θα περάσουμε τώρα στα άλλα μέλη της Επιτροπή μας. Uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με το ε, ερώτημα που αφορά τη διαδικασία. Για κάθε συνεδρίαση έχουμε μια συζήτηση περί της ημερησίας διατάξεως και υπάρχει ένας άγραφος νόμος που λέει ότι αν στο τέλος, αν δεν μπορείς να συμφωνήσεις για την ημερήσια διάταξη, το... ο οικοδεσπότης αποφασίζει για την ημερήσια διάταξη. Εμείς ε, καταστήσαμε σαφές ότι θα ήταν ε, καλύτερο να εστιάσουμε στο πεδίο και στο βαθμό της δραστηριότητας. Αλλά Πιστεύουμε πως είναι επίσης χρήσιμο να δούμε γενικά την εποπτεία, γιατί αυτό είναι τμήμα της ανέβρεσης στοιχείων ούτως ή άλλως. Τα έγγραφα που έχουμε ενώπιόν μας είναι δημόσια έγγραφα, τα οποία εμείς μελετούμε. Δεν λάβαμε έγγραφα από την κυβέρνηση των ΙΠΑ και δεν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε λεπτομερές πρόγραμμα δραστηριοτήτων, διότι μας είπαν ότι όλα αυτά είναι διαβαθμισμένα. Ζητήσαμε από τη ΣΥΠΑ να μας κάνουν έναν ε, ε, γύρο, μια ενημέρωση για τις ε, ε, Αυτό δεν κατέστη δυνατό δυστυχώς αυτή τη φορά. Την επόμενη συνεδρίαση φυσικά θα το ξαναζητήσουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι η σημασία της δραστηριότητας αυτού του δικαστηρίου για τις ΕΠΑ, ιδιαίτερα όσον αφορά το άρθρο 702 και τις δραστηριότητες εποπτείας. Η έρευνά μας έχει δείξει πως υπάρχει ε, ε, σχέση με το άρθρο 702 και βεβαίως ως τμήμα της ανέβρεσης στοιχείων θα ζητήσουμε από τους Αμερικανούς συναδέλφους να κατανοήσουμε καλύτερα την σχετικότητα αυτών των αποφάσεων από τη στιγμή που αυτά αφορούν στοιχεία προστασίας, αυτές μάλλον αφορούν στοιχεία προστασίας για τους πολίτες της Ένωσης. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα του κύριου Μωράης, επανειλημμένως έχουμε ζητήσει από την Αμερικανική κυβέρνηση να μας δώσει τουλάχιστον κάποιους άξονες για το πώς οι πολίτες επηρεάζονται στην Ένωση και πώς. Αναφερθήκαμε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ έχει δημοσιεύσει ένα ποσοστό ε, ε, κυκλοφορία στο ίντερνετ. Επιστήσαμε την προσοχή ότι ε, στο γεγονός ότι δεν θα πρέπει να είναι τεχνικός πολύ δύσκολο, ας πούμε σε σχέση με τα μεταδεδομένα και τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τουλάχιστον να μας δώσουν ένα χοντρικό νούμερο για το πώς ευρωπαϊκά τηλεφωνικά νούμερα έχουν ε, έχουν καταγραφεί για ανθρώπους που καλούν την ΣΥΠΑ ή καλούν ε, την Ευρώπη από τη ΣΥΠΑ. Το, καταστήσαμε σαφές πως είναι σημαντικό για μας να κατανοήσουμε τον αντίκτυπο της πρόσβασης στη, ε, στα υπερατλαντικά καλώδια, όπως φαίνεται να γίνεται, για τους πολίτες της Ένωσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμιά ένδειξη ως προς αυτό όσον αφορά την επιβεβαίωση των δραστηριοτήτων και των προγραμμάτων, τα μετα... η συλλογή χίδιν στοιχείων μεταδεδομένων ε, έχει επιβεβαιωθεί. Επίσης έχει επιβεβαιωθεί ότι το άρθρο 702 είναι η νομική βάση για το πρόγραμμα Πρίσμα. Αυτό το άρθρο μας ε, επεξηγήθηκε ως ένα στοχευμένο πρόγραμμα, αλλά η ευρύτερη συλλογή όλων όσων περνούν από το διατλαντικό καλώδιο δεν έχει επικυρωθεί ούτε έχει ε, υπάρξει άρνηση. Εμείς έχουμε υποδείξει στις ΕΠΑ ότι οι παρουσιάσεις για την εποπτεία είναι σημαντικές, αλλά για να καταλάβουμε τον αντίκτυπο στους Ευρωπαίους πολίτες πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο στο τι είναι νόμιμο σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία. Διότι η ανησυχία δεν είναι ότι παράνομα κατασκοπεύουν ε, τους Ευρωπαίους πολίτες σύμφωνα με την Αμερικανική, τον, Αμερικανικό νόμο, αλλά καταστήσαμε σαφές ότι η δική μας ε, μέρημνα είναι να δούμε τι είναι νόμιμο και τι όχι. Είπαμε λοιπόν ότι θέλουμε να έχουμε περισσότερη σαφήνεια για την ύπαρξη και τον αντίκτυπο των δραστηριότητα που σχετίζεται με την ε, συλλογή ε, μέσω του ε, περασλαντικού καλωδίου καθώς και στοιχείων που αφορούν εταιρείε και ιδιαίτερα το γι' αυτό το εξηγήσαμε στους Αμερικανούς συναδέλφους επειδή πολλά από τα στοιχεία που περνάνε από το καλώδιο δεν είναι διεθνείς επικοινωνίες με τις ΗΠΑ αλλά είναι εγχώριες εσωτερικές επικοινωνίες και αυτό το έχουμε πει επανελειμμένως. Ας στείλεις ένα SMS εγώ να στείλω σε εσά ένα μήνυμα που λέει τι γίνεται, ενώ είναι τελείως ενδοευρωπαϊκή επικοινωνία, τα στοιχεία περνάνε από το καλώδιο και φτάνουν κατευθείαν στη ΣΥΠΑ. Αν ε, ρωτήσεις μια ερώτηση σε κάποιο ε, site του Google, του Google πάλι περνά αυτόματα στην Καλιφόρνια. Ε, Αυτές τις ερωτήσεις λοιπόν τις έχουμε θέσει, αλλά δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Το πεδίο της συζήτησης είπαμε ότι είναι ανέβρεση στοιχείων και γι' αυτό δεν έχουμε μπει σε συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του ασφαλούς λιμένα, αλλά βεβαίως έχουμε επιστήσει στην προσοχή της κυβέρνησης αλλά και των δύο σωμάτων της σημασίας των αποφάσεων περί ασφαλούς λιμένα στο πλαίσιο αυτό και πιστεύω ότι αυτό που σαφώς διεφάνει είναι μια ανησυχία που τώρα έχει μεγαλώσει λόγω των όσων ακούμε για το SWIFT ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι μια, ένα σχήμα, ένα ε, σχήματο συμφωνιών ε, διμερών, οι οποίες όμως μετά υπονομεύονται από μονομερείς δραστηριότητες. Η ερώτηση του κυρίου Άλμπρεχτ. Ποια είναι η εκτίμησή μας όσον αφορά τις αλλαγές. Υπάρχει καμιά πολιτική βούληση για υπέρ των αλλαγών. Για να απαντήσω και εμέσως προς την κυρία Ιντιβέλτ, βεβαίω είμαστε ε, δημόσιοι υπάλληλοι και ενεργούμε κατόπιν εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με εκπροσώπους των 100 μελών που έχουν οριστεί από το Συμβούλιο, αλλά ο διάλογος πολιτικός βεβαίως και έχει ξεκινήσει και γίνεται ανάμεσα στον Αντιπρόεδρο και τον κύριο Χόλτερ. Εμείς είμαστε απλώ υπάλληλοι μπορείτε να είστε βέβαιοι ότι η ίδια η Αντιπρόεδρος όχι μόνο ξεκίνησε, αλλά ε, είναι απόλυτα δεσμευμένη σε αυτή τη δραστηριότητα. Τώρα, το γεγονός ότι δύο σώματα έχουν ερωτηθεί από τον Πρόεδρο για να υποβάλουν προτάσεις για πιθανές αλλαγές και για εκτίμηση της κατάστασης αποτελεί ένδειξη ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την ανέβρεση πιθανών κινήσεων εναλλακτικών επιλογών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας επίσης μάθαμε ότι η Αμερικανική βιομηχανία όλο ένα και πιο ξεκάθαρα μιλά προς το κοινό και προς το Κογκρέσο για τη ζημιά που έχουν προκαλέσει αυτοί οι ισχυρισμοί ε, παγκοσμίω για τις επιχειρήσεις τους. Και θα έλεγα ότι η συζήτηση συνεχίζεται. Είναι μια συζήτηση που εν μέρη αφορά τις ε, θέματα πολιτικών ελευθεριών ίσως είναι και το πιο σημαντικό τμήμα τη συζήτηση, και έπειτα υπάρχει και μια αναδυόμενη συζήτηση για τον διεθνή οικονομικό αντίκτυπο όλων αυτών και υπάρχουν ορισμένοι Αμερικανοί, αμερικανικοί ενδιαφερόμενοι φορείς που υψώνουν τη φωνή τους προς το συμφέρον των λαών εκτός των ΗΠΑ ε, για το ποιον τα θεμελιώδη δικαιώματα θίγονται από αυτές τις δραστηριότητες και φυσικά κάθε φορά που ακούμε ε, υψωμένη τη φωνή των λαών είμαστε πολύ ευγνώμονες γιατί δεν γίνεται συχνά κάτι τέτοιο. Μελετούμε όντως τις ε, γνωμοδοτήσεις ε, του δικαστηρίου Pfizer που είναι δημοσιευμένες. Ε, βλέπουμε ε, σε εξηγήσει ε, και τη σημασία των δραστηριοτήτων του δικαστηρίου αυτού και τις επιπτώσεις των αποφάσεών του για τους Ευρωπαίους πολίτες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του οικονομικής κατασκοπίας. Επανελειμμένως έχουμε λάβει προφορικός εγγυήσεις ότι σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία δεν είναι νόμιμο να γίνεται οικονομική κατασκοπία. Και αυτό ήταν το τμήμα της δήλωσης του Προέδρου Ομπάμα στην Σουηδία. Ωστόσο δεν λάβαμε τίποτα γραπτό ούτε σαφείς ενδείξεις για το πού αν αποκλείεται κάτι τέτοιο σύμφωνα με την νομοθεσία, σύμφωνα με ποιο νόμο είναι παράνομο. Και επίσης εξασφάλιση ότι οι, ότι ιδιώτες ε, σύμβουλοι που ανταγωνίζονται παγκοσμίω ε, και παρέχουν υπηρεσίες προς τη κοινότητα μυστικών υπηρεσιών των είπα ότι δεν χρησιμοποιούν αυτά τα στοιχεία για άλλους σκοπούς. Δεν έχουμε ακόμα λάβει οποιαδήποτε εξασφάλιση. Για το ποιοι δηλαδή είναι οι μηχανισμοί που προβλέπονται στη ΣΥΠΑ ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όμω έχει σημειωθεί το δικό μα ενδιαφέρον να γνωρίζουμε περισσότερα και ελπίζουμε ότι στο μέλλον, σε κάποια μελλοντική μας συνάντηση θα ενημερωθούμε για τα θέματα αυτά. Okay, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ίσως για το τελευταίο που είπατε, σε απάντηση στη ερώτηση του Άξελ Φως, θα μπορούσαμε ενδεχομένω να ρωτήσουμε και άλλου επιτρόπου, ε, του αρμοδίου για τα θέματα του ανταγωνισμού ή εμπορίου ενδεχομένω. Θα του ενδιαφέρουν, φαντάζομαι. Έχω δύο συναδέλφου ε, ε, που θέλουν το λόγο και κάποιοι άλλοι. I think that's it. Mrs. If you could... Κυρία Ζήπελ, ναι και την κυρία Μαγκάτη σημείωσα. Δύο λεπτά ο καθένας το πολύ παρακαλώ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Θέλω να σταθώ σε δύο τομείς μονάχα. Στην τελευταία συνάντησή μας είχαμε ασχοληθεί με το θέμα της εποπτείας και είχε φανεί ότι το θέμα του, της έκτασης της ε, συλλογής δεδομένων ήταν και αυτό ένα σημαντικό θέμα, μέχρι που εκτείνεται δηλαδή η συλλογή πληροφοριών. αναφέρθηκε ότι θα μπορούσαν να ανασφορέσουν να εξασφαλίσει την προστασία της προσωπικής ζωής, αλλά το ερώτημα ήταν αν υπάρχουν σκέψεις στις Ηνωμένε Πολιτείε πώς θα μπορούσε αυτή η άκρητη συλλογή δεδομένων στρατηγικού χαρακτήρα να περιοριστεί και κατά πόσο η Κομισιόν θα ήταν σε θέση να δώσει κάποιες κατευθύνσεις στους Αμερικανούς για, να, για το πώς θα έπρεπε να πράττουν. είναι καλό να ξέρουμε το αν είναι κάτι ε, με τους δικούς μας κανόνες, μάλλον ότι είναι με τους αμερικάνικους κανόνες νόμιμο ή όχι, χρήσιμο είναι, αλλά το θέμα είναι πιο σημαντικό για μας ως ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου, το κατά πόσο συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με αυτές τις ε, ε θέσεις των Αμερικανών. Επίσης, για το θέμα της ε, οικονομικής κατασκοπίας είναι σαφές ότι ακόμα και η NSA βλέπει να υπάρχει μια διαπλοκή ιδιωτικών και δημοσίων συμφέρον, συμφερόντων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να σκεφτούμε για νέους κανόνες, γιατί αλλιώς τελικά βλέπουμε ότι ένα μεγάλο μέρος της επεξεργασίας γίνεται από επιχείρηση και αυτό αποβαίνει σε βάρος των δικών μας επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Ένα τελευταίο ερώτημα προς τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Είδαμε σε κάποια δημοσίευση στις Ηνωμένες, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια στιγμή μονάχα, ότι ένα μεγάλο μέρος της όλης διαδικασίας ξεκινάει από οικονομικά συμφέροντα. Και θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στοιχεία που να επιβεβαιώνει ή όχι αυτή τη θέση. Και εγώ συνεχίζω αυτά που είπε η συνάδελφος η κυρία Ζίπελ. Εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πολλές ουσιαστικές πληροφορίες. Εμείς θα πρέπει να περατώσουμε βέβαια τη σύνταξη της ε, εκθέσεως για φέτος. Δεν έχουμε τώρα μια επαρκή επισκόπηση της κατάστασης και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από μια επιφανειακή επισκόπηση μοναχά. Δεν μπορούμε να μπούμε στις ε, ε, λεπτομέρειες. Δεν ξέρω αν αυτό θα αλλάξει. Δεύτερο, ο κύριος Μωράης έθεσε το ερώτημα της το ποσοτικό, δηλαδή τι έχει προέλθει από αυτή την επισκόπηση πόσους ε, αφορά και το θέμα της ποιότητάς τους. Επίσης υπάρχει ένα ακόμα πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι οι Αμερικανοί έχουν μια διαφορετική αντίληψη του προβλήματος από ότι εμείς. Μας είπαν ότι οι Αμερικανοί έχουν ένα κάποιο ανοιχτό πνεύμα για αλλαγή, ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσει για την εξωτερική της πολιτική. Όλα αυτά δεν νομίζω ότι μας ικανοποιούν θα θέλαμε να ξέρουμε καλύτερα τι δυνατότητες υπάρχουν για όλα αυτά. Ο κύριος Μπρόνς. Είπε ο κύριος Ζέλε ότι υπήρχαν μορφές υποπτίας που εξετάζαν κατά πόσο είναι σύμμορφη με το αμερικανικό δίκαιο αυτή η παρακολούθηση και εάν έχει νόημα σε επίπεδο πολιτικό. Οι μόνοι οι οποίοι ασχολούνται με όλα αυτά τα θέματα σε επίπεδο νομικό είναι οι Ευρωπαίοι και οι τρίτε χώρε. Αλλά οι Αμερικανοί είναι φανερό ότι θεωρούν ότι υπάρχει μόνο μια μορφή δικαίου που είναι το Αμερικάνικο δίκαιο και όλα τα άλλα είναι διάφορα ενοχλητικά έθιμα που ονομάζουν νόμου οι υπόλοιποι στον κόσμο. Ένα μεγάλο μέρο αυτή τη παρακολούθηση έχει γίνει με το να χρησιμοποιεί τεχνολογία για να παρακαμφθούν οι διασφαλίσεις που προβλέπονται από αυτή τη συμφωνία. Επομένω, οποιαδήποτε συμφωνία ή αλλαγή τη συμφωνία δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα γιατί οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να ε, ανακόψουν και να ελέγξουν όλες τις πληροφορίες που περνάνε από τις Πολιτείε. Λοιπόν, ακόμα και αν υπήρχε μια συμφωνία, η αρμόδια εταιρεία μπορεί να συνεχίσει να κάνει την παρακολούθηση ανεξέλεγκτη. Το μόνο το οποίο μπορεί να περιμένει κανείς είναι αν υπάρξει μια αντίδραση στι ΗΠΑ για αυτή την παρακολούθηση. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει κάτι από την ίδια την NSA. Κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ. Δεν άκουσα δυστυχώ τα πρώτο μέρο των σχολείων του κυρίου Νέμιτσα. Συγγνώμη γι' αυτό. Τέλο πάντων, θα μπορούσατε να μα πείτε αν σα εξέπληξε αναγνώριση από το Υπουργείο Οικονομικών των είπα παντώντα στην ε, Επίτροπο Μάλστρομ. Βέβαια είστε σε άλλη γαματέλτα, αλλά τέλο πάντων. Συγκεκριμένα σε εσά από τη γαματέλτα Jazz, θέλω να ρωτήσω. Σα εξέπληξε η αναγνώριση από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για τα δεδομένα SWIFT, ότι δηλαδή αποκτώνται εκτό του πλαισίου τη συμφωνία TFTP. Αυτά τα λέει ο κύριο Κόεν στην απάντησή του. Αναφέρεται επίσης σε κλητεύσεις, σε δικασίες κλητεύσεις. Τώρα δεν ξέρω ε, αν αυτό αφορά το SWIFT το ίδιο ή με μονομένους χρηματοψηφικούς οργανισμούς. Πάντως αναφέρεται το θέμα αυτό. Και βέβαια δεν μας εκπλήσει το ότι δεν λένε τίποτα σε σχέση με το κατά πόσον ε, τις αναχαιτήσεις ή τη, τα στοιχεία που συλλέγονται από την NSA τα συμπεριλαμβάνουν ή όχι. Αυτό εσείς θα το λέγατε παραβίαση της συμφωνίας SWIFT. Δηλαδή αν ε, υπήρχαν ε, συνεχώς ε, εντολές, εντάλματα, κλητεύσεις για την παροχή δεδομένων στο πέσο του SWIFT. Ή τα περιλαμβάνει όλα το εσείς κατά την άποψή σας. Και αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη βοηθητική τέτοια διαδικασία. Και αν το NSA ή άλλη η υπηρεσία είχε άμεση πρόσβαση. Αυτό είναι εκτός πλαισίου Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, άρα δεν αφορά καθόλου ε, και δεν λαμβάνεται υπόψη το, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού δεν καλύπτονται, δεν περιλαμβάνει, δεν διέπει αν θέλετε τις υπηρεσίες πληροφοριών. Κυρία Μορβάη, ευχαριστώ πολύ. Ούτε εγώ άκουσα την αρχή της παρουσίασης του κυρίου Νέμιτς. Τέλος πάντων, ε, μεταξύ 2 και 3 Υπήρχε ένα πρόγραμμα, είχαμε εκφράσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, επικρίσεις κατά του Αζερμπαϊτζάν ε, που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπήρχε κάτι τραγιλαφικό και κομικοτραγικό που συνέβαινε. Δηλαδή ότι αυτό το γεγονός, αυτό το συμβάν έγινε ε, όσο είχε διάλειμμα αυτή η Επιτροπή. Τέλο δεν θα μπούμε σε όλε τι λεπτομέρειε για νομοθεσία είπα, ούτε για την ομολογία των Αμερικανικών δικαστηρίων σε σχέση με υποθέσεις που αφορούν ε, επικόους ε, ευρωπαϊκών χωρών που τους υπέκλεψαν τα στοιχεία τους. Εγώ είμαι νομικός και βλέπω πολύ περίεργα πράγματα να συμβαίνουν. Λάβαμε ένα έγγραφο Έχουμε και το κανονισμό ΦΙΣΑ. Στο 2021 21 λέει ότι όταν υπάρχει συλλογή δεδομένων μπορεί κάποια από αυτά τα στοιχεία να είναι χρήσιμα κάποια στιγμή για την, ε, τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας, άρα είναι αποδεκτό να διατηρούνται αυτά τα δεδομένα. Μπορεί να είναι αποδεκτό αυτό σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία, αλλά εμείς εδώ μιλάμε και για το ευρωπαϊκό δίκαιο. Μπορεί να έχουμε κάποιες μορφές πορνογραφίας, παιδικής πορνογραφίας, για παράδειγμα, που είναι αποδεκτές στη ΣΥΠΑ. Δεν ισχύει το ίδιο στην Ευρώπη. Πρέπει να σωτευτούν τα παιδιά. Άρα αυτό που θέλω να πω εν κατακλείδη είναι ότι μπορεί κάτι να είναι αποδεκτό στις Ηνωμένε Πολιτείε ή νόμιμο, γιατί τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα. Ε, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεχθούμε εμείς αυτή την ε, θεώρηση. Εμείς πρέπει να είμαστε κατά και πρέπει να προσπίσουμε τα ε, θύματα. Ναι, είμαστε αιρετοί εκπρόσωποι και γνωρίζουμε τι κάνουν οι κυβερνήσεις μας. Αν οι Αμερικανοί είναι φίλοι μας, θα πρέπει να γνωρίζουμε και το τι κάνει η κυβέρνησή τους. Δεν νομίζω πως σε μια δήλωση που λέει ότι απλώς αυτό που κάνουμε είναι νόμιμο αρκεί. Θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Και αυτοί οι άνθρωποι της εποπτείας δεν τους εμπιστευόμαστε πλέον. Μόνο αν γνωρίζουμε για ποιο λόγο χρησιμοποιούν το νομοθεσία μπορούμε να κρίνουμε για να δούμε αν αυτό που κάνουν νόμιμο ή όχι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά το εμπορικό απόρριτο. Μας λένε να μην ανησυχείτε ή απαγορεύετε. Άμα διαβάσετε την παράγραφο 1883 του δικού τους ε, κώδικα, λέει ότι εδώ δεν εμποδίζεται καμιά άλλη νομίμη διαδικασία που, ε, στην οποία προβαίνει η κυβέρνηση. Άρα η κυβέρνηση εξαιρείται. Τι ε, αξία έχει μια προφορική δήλωση λοιπόν. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών και θα ζητήσω από τον κύριο Νέμιτς να απαντήσει. Έχω και ένα στοιχείο που αναφέρατε ότι το στο είναι τα μέλη μάλλον του Κογκρέσου συμμετέχουν επίσης σε αυτές τις συνόδους. Ε, είναι όντως αλήθεια ή όχι. Ναι, για την τελευταία ερώτηση, Πρόεδρε. Έχουμε συναντήσει χωριστά στο Κογκρέσο υπαλλήλου ε, της, Επο... της Επιτροπής ε, Εποπτείας της Γερουσίας για μια ώρα για ανταλλαγή απόψεων, αλλά δεν συμμετέχουν στις συζητήσεις ε, κυβέρνησης, της κυβέρνησης προς εμάς, με εμάς. Για τα θέματα περιορισμού για, τη στρατηγική υποπτία και χωρίς καμιά υποψία. Δηλαδή το θέμα των ε, ε καλωδίων. Το πρώτο θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τίποτα παραπάνω από τις συζητήσεις μας με τη για το τι ακριβώς γίνεται ή δεν γίνεται. Δεν έχουν επιβεβαιώσει ούτε έχουν αρνηθεί το ότι παίρνουν στοιχεία από το, τα υπερατλαντικά καλώδια. Ενδιαφερόμαστε γι' αυτό που αυτό υποκαλούν το νόμο καλών πρακτικών περιποπτείας και με μεγάλο υπερηφάνεια ήθελα να μας το παρουσιάσουν με έναν εντυπωσιακό αριθμό. Δεν ήθελα να δώσω ε, ε, ποιοτική κρίση, αλλά υπάρχει ένας εντυπωσιακό αριθμός σωμάτων εποπτείας στο Υπουργείο Εθνικής ε, ε, κατασκοπίας μέσα στο, μέσα στο έχουν 30 ε, υπαλλήλου για την Επιτροπή Εποπτείας ε, και λάβαμε και μια σύγκριση της οποίας την ακρίβεια δεν έχουμε ελέγξει για τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη σε μια προσπάθεια να αποτραπεί η δραστηριότητα αναζήτησης ε, στοιχείων στην ουσία μας επιστρέφουν την ερώτηση ε, και μας λένε εσείς τι κάνατε ακριβώς. Εμείς απαντούμε λοιπόν ε, ως εξή. Αν θέλετε να δείτε τους περιορισμούς της εποπτείας από τις μυστικές υπηρεσίες χωρίς καμιά υποψία, παρακαλώ διαβάστε την νομοθεσία των κρατών μελών μας και θα βρείτε πολύ καλά παραδείγματα και λιγότερο καλά. Αλλά θα δείτε παραδείγματα που περιορίζουν αυτού του είδους τη δραστηριότητα πολύ πιο αυστηρά από ό,τι φαίνεται να περιορίζονται στη, σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία και το τονίσαμε αυτό στους συναδέλφους των ΕΠΑ. Για το θέμα της ε, ιδιωτικής συμμετοχής ή όχι, εμπλοκής ή όχι, δεν έχουμε συζητήσει παρά Ζητάμε στοιχεία, ζητάμε διευκρινήσει. Πώ, α πούμε, εξασφαλίζει η Αμερικανική κυβέρνηση ότι οι στοιχεία ιδιωτική ίση που συλλέγονται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων υποπτία δεν χρησιμοποιούνται από του ε, ιδιώτε ε, συνεργάτε για άλλου σκοπού. Επίση, ρωτήσατε τώρα για το χρονικό πλαίσιο. Η ΕΠΑ προσέφεραν μια επόμενη συνάντηση σε επόμενε εβδομάδε. Δεν έχει ακόμα καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Ελπίζουμε πω θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε πολλά από τα θέματα που κι εσεί αναφέρατε εδώ, δηλαδή το πεδίο εφαρμογή των δραστηριοτήτων, πώ οι Ευρωπαίοι ε, μπλέκονται, ποιοι είναι οι περιορισμοί, γιατί, αυτές, γιατί στοχεύονται αυτοί οι Ευρωπαίοι και γιατί, εν πάση περιπτώσει, συλλέγονται τα στοιχεία του για ποιου σκοπού. Ελπίζουμε επίση πω θα μπορέσουμε να δούμε και την άλλη πλευρά του νομίσματο τη να δούμε δηλαδή πόσο επιτυχή είναι αυτά τα προγράμματα. Έχουμε, βάλει, έχουμε θέσει πολλέ ερωτήσει, αλλά δεν έχουμε πάρει καμιά παραπάνω απάντηση από αυτά που βλέπουμε και στι εφημερίδε. Τώρα, μετά από την επόμενη αυτή συνεδρίαση θα πρέπει να δούμε ποια θα είναι η κατάσταση, αλλά η Κομισιόν σκοπεύει να κάνει γραπτή αναφορά πριν το τέλος του έτους. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις για πολλά ζητήματα, όπως η έμφαση στην εποπτεία, μας έδειξε ότι είπα στην ουσία έχουν ως σημείο αναφορά στον εαυτό τους. Το πιο σημαντικό θέμα είναι κατά πόσο κάτι τέτοιο είναι νόμιμο για την Αμερικανική νομοθεσία. Ε, τα ακούσαμε αυτά με ευγενικά βέβαια αυτή τη φορά, αλλά τους καταστήσαμε σαφές ότι δεν μας ενδιαφέρει αν είναι νόμιμο όλα αυτά ε, σύμφωνα με την Αμερικανική νομοθεσία, αλλά το ότι όλοι οι πολίτες μας έχουν θεμελιώδη δικαιώματα και θέλουμε τα δικά τους δικαιώματα να προστατεύονται και γι' αυτό και θέλουμε να κατανοήσουμε το πεδίο των δραστηριοτήτων των ΙΠΑ γιατί μπορεί αυτές να παραβαίνουν το δικαίωμα τα δικαιώματα μάλλον των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό το έχουμε επανειλημμένως ε, δηλώσει. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του TFTP που έθεσε η κυρία Λότφορντα θα ήθελα να παραπέμψω την ερώτηση στο συνάδελφο Πρίμπε που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια. Έχουν και... Um, Ευχαριστώ πολύ. Εν συντομία, γιατί το θέμα αυτό έχει συζητηθεί με πολύ λεπτομέρεια σήμερα το πρωί, να προσθέσω στις ε, πληροφορίες που σας δόθηκαν ότι και αυτή η ομάδα ad hoc εξέφρασε τις ανησυχίες της για τις καταγγελίες για το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλοι διάβλοι πλέον της TFTP για τη μετάδοση δεδομένων. Και αυτό το αναφέραμε λοιπόν στη διαβούλευση που γίνεται. Φυσικά συνδέεται αυτή με τη γενικότερη συζήτηση που έχουμε στην ομάδα ad hoc. Όπως είπε και η Επίτροπος Μάλιστον σήμερα το πρωί. Έχουμε κάποια ερωτήματα για την επιστολή του κ. Κοέν και είναι ακριβώς αυτά τα ερωτήματα που μας έχετε θέσει εσείς και που πρέπει να διασαφινιστούν. Δεν μπορείτε να περιμένετε από μένα να σας πω περισσότερα γιατί συνεχίζεται αυτή η διαδικασία. Επιτρέψτε μου. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι καταγγελίες ευσταθούν κατά τη δική σας άποψη, εσείς είσαστε νοματής, αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας. Ακόμα περισσότερο η οχι τη συμφωνιας ακομα περισσοτερο η επιστολη του κυρίου Κοέν δεν λέω ότι παραδέχεται, αλλά αναγνωρίζει με σαφή τρόπο ότι, τα δεδομένα, ότι κάποια δεδομένα του SWIFT συλλέγονται έξω από το πλαίσιο του TFTP. Εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο, είναι παραβίαση ή όχι. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Νέμιτς. Είναι η συνολική άποψη της Κομισιόν ότι είναι έτσι. Τώρα ποιος θα απαντήσει, αυτό είναι δικό σας θέμα. Θα ήταν, μια, μια παραβίαση ή όχι κάτι τέτοιο. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα κυρία Λάτφορτ. Όπως ελέγχεται την Επίτροπο ε, Μάστον, αυτό θα πρέπει να είναι το αντικείμενο περαιτέρω διαβουλεύσεων. Όχι, δεν κατάλαβα το ερώτημα. Το ερώτημα είναι εάν κάποιος εισβάλλει σε ένα μαγαζί. Θεωρείται αυτό ότι είναι Διάρεξη η νομική σας άποψη. Δεν περιμένουμε να μας πείτε αν είναι σωστές ή όχι αυτές οι καταγγελίες. Αν αληθεύουν, αν συλλέγονται δεδομένα εκτός της συμφωνίας TFTP, κατά τη δική σας άποψη, είναι αυτό παραβίαση της συμφωνίας ή ου. Αν κάποιος μπει σε ένα μαγαζί είναι διάρρηξη. Αν οι Αμερικανοί έχουν παραβιάσει τη συμφωνία, αυτό θα διασαφινιστεί στι διαβουλεύσει. Ευχαριστώ που δεν απαντάτε το ερώτημα. Κάντε μία δήλωση, η Κομισιόν δεν απαντάει την, στην ερώτησή σα. Θέλετε να απαντήσετε στα άλλα ερωτήματα, κύριε Νέμιτ. Νομίζω τα άλλα ερωτήματα δεν ήταν ερωτήματα, ήταν δηλώσεις. Δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει να απαντήσω σε κάποιο ερώτημα. Πετε μου ποιο ερώτημα δεν απήντησα. No, no, I just clarify what maybe was not... Να διευκρινίσω, ίσως δεν καταλάβατε ότι αυτό είναι ερώτημα για την οικονομική κατασκοπία. Τι εγγυήσει μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί ότι δεν κάνουν οικονομική κατασκοπία. Με ποιο τρόπο οι πληροφορίε που συλλέγονται δεν χρησιμοποιούνται. Πώ θα εξασφαλίσουμε ότι χρησιμοποιούνται πληροφορίε για οικονομική κατασκοπία. Η απάντηση είναι δεν έχουμε καμία εγγύηση για αυτό το θέμα. Έχουμε πάρει επίσημε δηλώσει από τον πρόεδρο Ομπάμα ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν το κάνει. Αλλά δεν μας έχουν διευκρινίσει αν αυτό αποκλείεται από το νομικό σύστημα των ΗΠΑ και ποια είναι τα νομικά συστήματα τα οποία εξασφαλίζουν ότι οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες αναλύουν αυτά τα δεδομένα δεν τα χρησιμοποιούν για άλλους σκοπούς. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν πολύ σαφές. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Νομίζω θα τα ξαναπούμε. Ερχόμαστε λοιπόν στην τρίτη ανταλλαγή απόψεων. Ανταλλαγή απόψεων με την κοινωνία των πολιτών στις ΗΠΑ. Ξεκινάμε με τον κύριο Γέπεσεν, ο οποίος είναι ο Διευθυντής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοκρατίας και Τεχνολογίας. Θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση. Δυστυχώς ο πρόεδρος του κέντρου, αυτού ο κύριος, η κυρία Λέσλι Χάρις, δεν μπορεί να είναι παρούσα γιατί είχε ένα μικρό ατύχημα και δεν μπορούσε να είναι εδώ. Της ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση. ανάρρωση. Και μετά ο κύριος Νότζεϊμ από το project για free, Project for Freedom, Security and Technology αυτού του κέντρου θα απευθυνθεί σε εμά μέσω βίντεο διάσκεψης και μετά θα μπορέσουμε να κάνουμε ερωτήσεις αμφί και στους δύο αυτούς κυρίους. Ο κύριος Γέπεσεν πρώτα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την εισήγηση που κάνατε. Με μεγάλη χαρά συμμετέχουμε στην έρευνά σας και σας συγχαίρουμε που συστήσατε αυτή την ερευνητική ε, είναι η μόνη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην, ε, στην Ευρώπη. Κανένα εθνικό κοινοβούλιο δεν προέβησε τέτοιο βήμα. Καταρχήν το Κέντρο για τη Δημοκρατία και την Τεχνολογία να σας πω ότι είναι, είναι μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών με στόχο την υπεράσπιση των πολιτικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο ψηφιακό περιβάλλον. Ε, είμαστε φωσιωμένοι στο να είναι ανοιχτό, δημοκρατικό και δωρεάν το ίντερνετ. Ε, είναι μια... Στις ΕΠΑ βοηθήσαμε να, να, να, να γίνει αντίσταση στο, στο Patriot Act και στο Peace Amendments Act και έχουμε οργανώσει μια μεγάλη, ένα μεγάλο συνασπισμό στο Αμερικανικό Κογκρέσο καλώντας τους πολιτικούς να ενισχύσουν την προστασία του, της ιδιωτικότητας ε, μέσα στο, μέσω του νόμου περί ιδιωτικού χώρου στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ε, για αυτή την έρευνα γίνεται μια αναθεώρηση της προστασίας ε, έναντι της ε, εποπτείας για πολίτες και μη πολίτες και κυρίως τα κενά που υπάρχουν στην προστασία αυτή Έπειτα προσφέραμε μια ανάλυση των βασικών προγραμμάτων εποπτείας που έχουν αποκαλυφθεί ε, για τη συλλογή στοιχείων σύμφωνα με το τμήμα 2.15 του Patriot Act, κυρίως για τη συλλογή στοιχείων μη ε, ε, πολιτών μετά την τροποποίησή του το 2008. Στη συνέχεια βλέπουμε τα αιτήματα της κοινωνίας των πολιτών για μεταρρύθμιση του νόμου περιποπτείας. Έχουμε κάποιες παρατηρήσεις για την κατάσταση στην Ευρώπη και ποια μέτρα θα μπορούσαν να ληφθούν διεθνώς ε, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις αποκαλύψεις η CDT συνεργάζεται με άλλες ομάδες, εταιρείες, υπερασπιστές, μέλη του Κογκρέσου για να επιτύχει τη μεταρρύθμιση των Αμερικανικών ε, προγραμμάτων εποπτείας από τον Ιούνιο. Για διάφορους λόγους, μεγάλο κομμάτι των πληροφοριών ρέει μέσω των ε, ΗΠΑ, διότι οι πάροχοι αποθηκεύουν στις ΗΠΑ πολλά από τα στοιχεία ε, Επιπλέον, οι ΙΠΑ έχουν αναπτύξει μοναδικές δυνατότητες για να κάνουν την εποπτεία και να συλλέγουν ε, στοιχεία από τα προϊόντα αυτής της εποπτείας. Με το επίπεδο δυνατοτήτων εποπτείας και πρόσβαση στα στοιχεία που έχουν οι ΙΠΑ, έχουν, φέρουν και αυξημένε ευθύνε. Είναι πιθανόν η NSA να κάνει τα προγραμματά τη με την πλήρη γνώση των, ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών, αλλά αυτό δεν ε, έρει τι ευθύνε τη αμερικανική κυβέρνηση, γιατί ε, πρέπει να προστατεύει όχι μόνο τα δικαιώματα των Αμερικανών, αλλά και των Ευρωπαίων και όλων παγκοσμίω. Και, και εμείς σε αυτό πιστεύουμε. Να συνοψίσω τι προτάσει που έχουμε υποβάλει. Πρώτον, ο, το, ο θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε ο νόμος να μην επιτρέπει στην NSA να συλλέγει χίδιν στοιχεία επικοινωνιών. Αντίθετα θα πρέπει να περιορίζονται σε αρχεία που αφορούν τερομοκράτε, κατασκόπου κτλ. και αυτού που έρχονται σε άμεση επαφή μαζί τους. Αθώε καθημερινέ επικοινωνίε ε, Αμερικανών πολιτών αλλά και όσων εκτός αμερική επικοινωνούν με τη ΣΥΠΑ να μην συλλέγονται χοντρικώ σε βάση δεδομένων που θα αναλύεται ανάλογα με το πότε θέλει η NSA. Χρειάζεται μεταρρύθμιση των διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες το δικαστήριο Φάιζα αναλύει και βγάζει τις αποφάσεις του. Είναι μυστικές οι διαδικασίες ε, του, του δικαστηρίου Φάισε και πολύ σπάνια μπορεί κανείς να δοκιμάσει αν στέκουν όλα αυτά σε ένα ανοιχτό δικαστήριο. Οπότε μπορεί κανείς να πει ότι όλα αυτά δεν είναι καν ε, μέσα στα πλαίσια της ε, ελευθερίας. Ε, η μυστικότητα γύρω από την εποπτεία θα πρέπει εν μέρη να αρθεί. Το, θα πρέπει να δοθεί επίσης η βάση ερμηνείας ε, του δικαστηρίου ΦΑΙΣΑ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να αποκαλύπτει τα αιτήματα εποπτείας ε, και επίσης τον αριθμό των ανθρώπων των οποίων αποκαλύπτονται οι πληροφορίες με βάση αυτήν την ε, άδεια από το δικαστήριο. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται η φύση και ο αριθμός των ετοιμάτων για στοιχεία και ο αντίκτυπος στους ε, πελάτες τους. Οι ΙΠΑ θα πρέπει να αναγνωρίσουν και να ε, ε, ε, προστατεύουν την ε, ιδιωτικότητα των Ευρωπαίων και άλλων σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι στιγμής δεν, έχει, δεν το έχει κάνει αυτό, ακόμα και αν το δικαίωμα σε, στον ιδιωτικό χώρο του άρθρου 17 του Διεθνού Συμφώνου για τα πολιτικά ε, δικαιώματα το έχει συνυπογράψει. Υπάρχουν διάφορα άλλα μέσα για τα, υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν δικαιολογείται αυτή η εποπτεία που στερεί τα δικαιώματα ιδιωτικότητας των ανθρώπων εκτός των ε, ΗΠΑ. Επίσης, υπάρχουν προβλήματα για τις εταιρείες που, συλλέγουν πληροφορίες ε, εξωτερικές, ακόμα και αν οι στόχοι δεν είναι ύποπτοι τρομοκράτες, ε, κατάσκοποι κτλ. Τόσο ευρέως ορίζονται αυτές οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν και οποιασδήποτε δραστηριότητες. Ας πούμε κάποια διαδήλωση κατά του ρατσισμού ε, επίση καλύπτονται και σχετίζονται όλα αυτά στις αμερικανικές εξωτερικές υποθέσεις και γι' αυτό και εμπίπτουν στους περιορισμούς που διάπουν αυτές τις, αυτή τη εποπτεία και αυτό πρέπει να αλλάξει στόχοι ευρύς που περιλαμβάνονται τώρα στο πρόγραμμα PRISM θα πρέπει να αλλάξουν. Ε, τέλος, το να γίνεται εποπτεία από την πίσω πόρτα θα πρέπει να τεθεί εκτός νόμου ε, δεν θα πρέπει να παρακάμπτονται η Αμερικανική νομοθεσία από την NSA, όταν αυτή δηλαδή παίρνει πληροφορίες από άλλες ε, ε, υπηρεσίες ε, πληροφοριών των ΙΠΑ, όταν δεν μπορεί να τις αποκτήσει από μόνη της. Το πρόβλημα λοιπόν της ηλεκτρονικής εποπτείας των πολιτών είναι παγκόσμιας φύσης σε αυτή την εποχή παγκοσμιοποιημένων επικοινωνιών και πρόσφατα ο Φρανκ Ρούλ, ειδικός εισηγητής για τις τηλεπικοινωνίες ε, κατέληξε στο συμπέρασμα πως είναι επίγουσα η ανάγκη να μεταρρυθμιστούν ε, οι σχετικές νομοθεσίες της ΣΥΠΑ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο γιατί πρέπει να βοηθήσουν και να ορίσουν ένα σύνολο κανόνων που να μπορούν να εφαρμοστούν παγκοσμίω. Κατά τη γνώμη μας αυτό μπορεί να γίνει αν τα θεσμικά όργανα ΕΠΑ και ΕΕ συνεργαστούν. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να ορίσουν τις δικές τους εποπτικές αρχές και να αναπτύξουν μια κοινή αντίληψη για το πώς θα πρέπει να εφαρμόζονται αυτές οι αρχές για την ε, εποπτεία για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ταυτόχρονα η Ευρώπη θα πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με τη ΣΥΠΑ και να αναζητήσει μια κοινή υπερατλαντική ε, συνεννόηση για αυτούς τους κανόνες σε εθνικό ε, πλαίσιο αλλά και σε διασυνοριακό πλαίσιο. Έτσι, θα έρθουν, ελπίζουμε, όλες οι αμφιβολίες για τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και όλο τον κόσμο και θα πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο. Η διαδικασία μεταρρύθμισης θα πρέπει να ξεκινήσει με τη διαφάνεια. Υπήρξαν εντυπωσιακέ αποκαλύψει όσον αφορά τη φύση και το βαθμό συστηματική παρακολούθηση κάποιων κρατών μελών τη Ένωση. Ακόμα όμω δεν ξέρουμε αρκετά για τι πρακτικέ που ακολουθούν οι ΗΠΑ. Είναι δύσκολο να καταλάβουμε και να επαληθεύσουμε σε ποιο βαθμό οι νόμοι οι ευρωπαϊκοί μπορούν να σταθούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα τελευταία χρόνια εμείς προσπαθούμε να συλλέξουμε τις νομοθεσίες ε, σε διάφορες χώρες και έχουμε βρει πως βασικά είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε τις πρακτικές γιατί οι σχετικές νομοθεσίες είναι αόριστες και οι κυβερνητικές ερμηνείες είναι είτε διαβαθμισμένες είτε και απόρριτες όπως τις είπα. Οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων ε, έχουν ε, τονίσει αυτά τα προβλήματα και ορισμένοι ευρωβουλευτές έχουν επικρίνει ότι σχεδόν ε, απόλυτη σιωπή έχει επικρατήσει από πλευρά των ευρωπαϊκών κρατών από τότε που ξέσπασε αυτή η ιστορία. Και η ΕΠΑ πολύ, πολύ απρόθυμοι είναι στο να ανοίξουν τις, τα χαρτιά τους. Η εθνική ασφάλεια ούτως ή άλλως ε, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Τον Η εθνική ασφάλεια δεν καλύπτεται από τις ε, ισχύουσες νομοθεσίες, οπότε μάλλον μόνο μέσω ενός ε, κανονισμού ή ενός περιοριστικού ε, μέτρου όσον αφορά την ροή πληροφοριών. Μόνο κάτι τέτοιο μπορεί να περιορίσει την NSA και τους Ευρωπαίους ομολόγους της να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που θέλουν. Ταυτόχρονα όμως ασκείται οικονομική και πολιτική πίεση στην Αμερικανική κυβέρνηση να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση την οποία σας περιέγραψα και το Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει να ασκεί αυτή την πίεση. Αλλά κατά βάση χρειάζεται η Αμερικανική κυβέρνηση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δεσμευτούν για μια περατλαντική διαδικασία ώστε να αναπτυχθεί συνολική συνένεση για τα κριτήρια που θα πρέπει να ισχύουν όσον αφορά την ε, εποπτεία και την ε, ε, εποπτεία των στοιχείων για την ασφάλεια. Πιστεύουμε πως είναι και εκείνη η ώρα για να αναπτυχθεί η διαφάνεια, η ανταναλογικότητα και ο έλεγχος σε αυτές τις πρακτικές ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ώστε να γίνονται σεβαστές οι αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις δύο επικράτειες. Δεν υπάρχει χρυσός κανόνας και δεν είναι εύκολο, αλλά ε, αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ανησυχίες. Εμείς προσβλέπουμε στη συνεργασία με αυτή την Επιτροπή και με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκρέγκ Νότζιμ, αν προφέρω καλά το όνομά σας, είναι στην οθόνη. Με ακούτε, ναι, σας ακούω, λέει ο κύριος Νότσιμ. Ωραία. Σας ακούμε και εμείς. Ε, ένα χαιρετισμό, λοιπόν, θερμό απευθύνουμε στην άλλη ε, πλευρά του σύρματος. Ο εισηγητής και οι σκιώδες ε, θα σας απευθύνουν τις ερωτήσεις που έχουν. Έπειτα θα απαντήσετε και θα ξεκινήσει μετά ένας δεύτερος γύρος. Φαίνεται ότι η σύνδεση είναι μια χαρά. Αν όμως υπάρξει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, μας το επισημαίνετε, σας παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτο ερώτημα, ή μάλλον πρώτα ερωτήματα από τον εισηγητή μας, τον κύριο Μωράης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ε, τον ε, κύριο Τζέπεσεν και εγώ μάλλον σκοτώνω το όνομά σας τέλος πάντων. Να σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Αυτή είναι η πρώτη φορά ε, με την κοινωνία των πολιτών. Θα έχουμε και άλλες ε, τέτοιες ε, ευκαιρίες, αλλά είναι σημαντικό τώρα να έχουμε έτσι μία πρώτη εικόνα για το πώς εσείς αντιλαμβάνεστε την κατάσταση. Κάνατε εσείς την παρουσίαση. Δεν ξέρω αν το συγκράτησαν, αλλά στην πρώτη σας φράση είπατε ότι είναι η μόνη ουσιαστική έρευνα στην Ευρώπη. διεθνικές έρευνες δεν υπήρξαν. Έτσι ξεκινήσατε μιλώντας για την έρευνα αυτή. Εγώ ελπίζω να κάνετε λάθος και να έχουν υπάρξει ε, κοινοβουλευτικές έρευνες στην Ευρώπη. Νομίζω ότι υπάρχουν πόσες δεν ξέρω, αλλά ε, ίσως ο γραμματέας μας γνωρίζει περισσότερα, αλλά δεν ξέρω αν, κάνω, αν έχω καταλάβει σωστά. Τέλος πάντων, ε, γίνονται έρευνε. Για εσά που προέρχεστε από την κοινότητα των πολιτών, που βλέπετε την Ευρώπη, βλέπετε και τι Ηνωμένε Πολιτείε, πώ αντιλαμβάνεστε τα πράγματα αυτέ οι έρευνε Μήπως δεν ε, έγιναν σε βάθος, ε, μήπως ήταν πάρα πολύ γρήγορες, αδύναμες, χωρίς να θέλω να βάλω στο στόμα σας βέβαια ε, λέξεις ή να σας επηρεάσω, αλλά ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Πιστεύετε ότι αυτό που βλέπετε, αν δεν είναι μακροσκελής το ερώτημά το πόρισμα, τα πόρισμα μια τέτοια έρευνα που βέβαια έχει τη, τα όρια τη, ε, γιατί θα λάβει πολλέ δευτερογενεί πληροφορίε και έχει περιορισμού, προφανεί περιορισμού ε, όσον αφορά την ε, απόπειρα να έχει πρόσβαση σε αυτή την κατάσταση και στι πληροφορίε από τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Και το δεύτερο είναι ότι εσεί βλέπετε και στην κατεύθυνση των ΗΠΑ, εμεί θα επισκεφτούμε τη ΣΥΠΑ τον Οκτώβριο. Το ερώτημά μου είναι εμείς πρέπει να γνωρίζουμε τι γίνεται σε ό,τι αφορά την άσκηση πιέσεων ε, στο Κογκρέσο. Τον Ιούλιο φαινόταν σε ό,τι αφορά δύο στις συνδιαλέξεις, ε, τα ε, σε ό,τι αφορά τα τηλέφωνα και για το ΦΑΙΣΑ υπήρχαν πιέσεις, ε, μειώθηκαν πολύ χρηματοδοτήσεις. Ε, τι ακριβώς συνέβη. Υπήρξαν και κάποιοι που ζήτησαν να λογοδοτήσει ίσως η NSA. Τι γίνεται τώρα. Αυτή η όθηση που είχε δοθεί τότε και υπήρξαν διάφορα νομοσχέδια για να υπάρχει ε, μεγαλύτερη ευθύνη από πλευράς NSA. Ε, υπάρχει ακόμη αυτή η όθηση, αυτό το momentum ή έχουν ξεφουσκώσει τα πράγματα. Αυτό είχα να ρωτήσω. Δεν ξέρω αν ε, θέλετε, Πρόεδρε, και εσείς να σταματήσω τώρα ή να υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι. Πρόεδρος, δεν βλέπω να υπάρχει κάποιος μέρος του ΕΛΚ. Δεν είναι εδώ ο κύριος Φως, ούτε και εγώ θα πω τελευταία στον κατάλογο, στο λόγο τώρα λοιπόν στον κύριο Άλμπρεχτ. Εγώ δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω πλήρως την παρουσίασή σας, γιατί μόλις ήρθα. Έχω ένα ερώτημα για τα θέματα της, ε, των υπηρεσιών πληροφοριών, των δομών τους, όταν πρόκειται για τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρείτε ότι εμπίπτουν αυτές, εμπλέκονται μέσα στο τωρινό μας πλαίσιο και στην ολοκληρωμένη μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ότι υπάρχουν υπηρεσίες πληροφοριών που κατασκοπεύουν και σπιουνάρουν πολίτες και εταιρείε άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μήπως θα μπορούσε να υπάρχει κάποια ελπίδα να ξεπεραστεί αυτό με το να συμφωνήσουμε πάνω σε γενικές αρχές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα για τις νομικές βάσεις, γιατί φυσικά η συνδίκη επιτρέπει δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών για λόγους εθνικής ασφάλειας. Και πιστεύετε ότι υπάρχει και κάποιο νομικό πλαίσιο, παραδείγματος χάρη, για την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και αν αυτό καλύπτει την ε, συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες σε θέματα συλλογής πληροφοριών. Ο κ. Κύρκοφ. Σας ευχαριστώ. Τώρα ξέρω γιατί δεν θέλω να είμαι στην πρώτη, στις πρώτες σειρές ενός ε, κινηματογράφου γιατί θα λουμπάγκο με το λαιμό μου. Καλημέρα λοιπόν στον ε, εκπρόσωπο από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον κύριο Γεπεσέν επίσης θα ήθελα να σας θέσω το εξή ερώτημα. Αλλά θέλω να κάνω και μία δήλωση σε σχέση με τη μαζική παρακολούθηση των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωρίς τις ηλεκτρονικές δυνατότητες και την τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί, η λαοκρατική δημοκρατία της Γερμανίας είχε μια από τις πιο αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης με τη στάζη για πολλά χρόνια στην Ευρώπη. Δεν είχαν τεχνολογία φουκαράδες, αλλά λόγω της έλλειψης δημοκρατίας εκεί, το σύστημα αυτό ήταν πάρα πολύ αποτελεσματικό στην παρακολούθηση. Και φοβάμαι ότι η ισορροπία μεταξύ προστασίας της ιδιωτικής ζωής των πολιτών και περιορισμού των εξουσιών του κράτους ενώ διατηρεί κανείς τις ελευθερίες των πολιτών, αυτό είναι δύσκολο και την προστασία τους. Το ερώτημα είναι τώρα εξή. Η τεχνολογία τώρα αυτή προχωράει με τεράστια ταχύτητα. Η συλλογή πληροφοριών, οι επικοινωνίες, όλα αυτά προωθούν. Κάθε εβδομάδα έχουμε και ένα καινούριο μαραφέτη το οποίο μπορεί να κάνει την διακόμιση πληροφοριών υπάρχει κάποιο σημείο όπου γίνεται απαραίτητο για μας να δούμε την ανάγκη περισσότερων ελέγχων για όλα αυτά ή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που ενώ προχωρούμε και ξέρουμε ότι και οι εγκληματίες και οι τρομοκράτες προχωρούν και αυτοί στην ίδια τεχνολογική καμπύλη. Έχουμε μια αύξηση στη δυνατότητα προστασία των πολιτών μας όσο αυξάνει και η δυνατότητα συλλογή πληροφοριών. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια ρευστή κατάσταση. Θα ήθελα ξέρω ποια είναι δική σας άποψη, κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Δύο ερωτήματα στον κύριο Γέπεσεν που προέρχονται από την παρουσίασή σας. Νομίζω ότι είναι λογικό αυτό το οποίο άκουσα σήμερα και έχω κάθε λόγο να παραμένω εδώ που είμαι. Είπατε δύο πράγματα. Μεταρρύθμιση των μυστικών υπηρεσιών. Αυτό είναι κάτι το οποίο απαιτείται. Της μορφής που έχουν οι μυστικές υπηρεσίες. Μήπως μπορείτε αυτό να το εξηγήσετε καλύτερα. Τι εννοείτε. Οι μυστικές υπηρεσίες είναι αυτό το οποίο είναι. Τι σημαίνει αυτό σε επίπεδο ελέγχου. Πώς λειτουργούν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές εποπτείας στις ΗΠΑ, πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η εποπτεία σας και τι προτάσεις έχετε να μας κάνετε για την περαιτέρω συζήτηση. Δίνω στον εαυτό μου το λόγο τώρα ως σκιώδη συζητητή για τους φιλελεύθερους. Ένα απλό ερώτημα και στους δυο σας. Εξετάζεται επίσης και την πτυχή των χρημάτων, δηλαδή ποιες είναι, ποια είναι τα κονδύλια του προπολογισμού τα οποία αφορούν τις παρακολουθήσεις, αν υπάρχουν μυστικοί προϋπολογισμοί, αν πληρώνει η Αμερικανική κυβέρνηση τις κυβερνήσεις πέραν του κόστους τους για τη συλλογή δεδομένων, αγοράζουν δεδομένα κυβερνήσεις. Ποιο είναι και το άχθος για τις εταιρείες που προέρχεται από αυτήν την ε, διαδικασία παρακολούθησης. Θα ήθελα να έχουμε και μια πληρέστερη εικόνα της οικονομικής διάστασης για όλα αυτά. Αλλά και ποιες είναι οι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εποφελούνται από αυτές τις πολιτικές, γιατί υπάρχουν εταιρείε οι οποίες εξειδικεύονται στην παρακολούθηση και στην κατασκοπία. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά θα θέλαμε να ξέρουμε πόσα λεφτά βγάζουν από αυτήν την ιστορία. Ίσως, κύριε, μπορεί να ζητήσουμε από τον κύριο Νόζεμ να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που θέλει και μετά να επαληθούμε σε εσά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με το πρώτο ερώτημα για το πώς έχουν μεταρρυθμίσει το Αμερικανικό Κογκρέσο Είχαμε πράγματι μια περίοδο δραστηριότητα τον Ιούλιο, κάπως ε, τα πράγματα ε, ηρέμησαν τον Αύγουστο, γιατί βέβαια ήταν σε διακοπές ε, το Κογκρέσο. Με την επάνωδο όμως των μελών του Κογκρέσου ξεκίνησε ξανά αυτή η δραστηριότητα και έχουμε τώρα τον πρόεδρο Τη Επιτροπή, τη Κασικής Επιτροπής της Γερουσίας που μιλά σε ένα συμβάν, σε μια εκδήλωση και εκεί θα ε, παρουσιάσει τι μεταρρυθμίσει που προτίθεται να κάνει στο σχετικό νόμο για την επιτήρηση. Θα γίνει και μια ακρόαση αρχές Οκτωβρίου σε ό,τι αφορά την μετάρρυθμιση τη ΦΑΙΣΑ και την πέμπτη στην εβδομάδα στη Γερουσία και στη συγκεκριμένη Επιτροπή Πληροφοριών θα γίνει μια νομοθετική ακρόαση. Αυτό σημαίνει ότι ε, μάλλον σύντομα θα δημοσιευθεί ένα νομοσχέδιο για τη μετάρρυθμιση της ΦΙΣΑ και πρέπει να σας πω ότι στις ΗΠΑ μεταρρυθμίσεις στον πατριωτικό νόμο έχουν προχωρήσει, είναι πιο εξελιγμένες ό,τι αφορά τις προτινόμενε μεταρρυθμίσεις, μάλλον σε σχέση με τις προτινόμενες μεταρρυθμίσεις ό,τι αφορά ε, τη, το τροποποιητικό νόμο τη ΦΥΣΑ και του νόμους περί ασφάλειας και επιτήρησης. Δεν είναι δηλαδή το νομοθετικό θεματολόγιο τόσο ανεπτυγμένο σε αυτό τον τομέα. Αν τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητούσαν να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις ακροάσεις, θα ήταν δύσκολο για κάποιο μέλος του Κογκρέσου να τους το αρνηθεί. Αυτή είναι μια επιλογή ενδεχομένως που πρέπει να εξετάσετε. Ένα άλλο ερώτημα ήταν το ακολουθήστε τα χρήματα, ποια ήταν δηλαδή τα οικονομικά κίνητρα για τις εταιρείες που εμπλέκονταν και ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την επιτήρηση, την παρακολούθηση των πληροφοριών. Εμείς δεν ξέραμε τίποτα για τέτοιον προϋπολογισμό μέχρι ότι είχαμε τις διάρκειες Snowden. Τα τελευταία χρόνια ο συνολικός αριθμός των δολαρίων που έχουν δαπανηθεί σε αυτό το τομέα πρόσφατα αποκαλύφθηκε και η κυβέρνηση θεωρούσε τα τελευταία 40 χρόνια ότι ακόμα και μόνο το συνολικό ποσό να δημοσιοποιείται, αυτό θα βοηθούσε τους τρομοκράτες. Όλα αυτά βασίζονται στα έγγραφα τελικά τα οποία ε, διέρευσαν από τον κύριο Σνόντεν και βλέπουμε ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα. Κάποια πηγαίνουν στις εταιρείε ε, των οποίων απαιτείται η βοήθεια από τη κυβέρνηση για αυτή την ε, παρακολούθηση. Τώρα κατά πόσον αυτές οι εταιρείε βγάζουν κέρδος, δεν κατέστη σαφέ τουλάχιστον εγώ στα ποσά που είδα. Και αν είναι επικερδές, ε, αυτό το ποσό είναι μικρό. Δεδομένου το μεγέθο των εταιριών, ε, τα ποσά είναι μικρά ω κέρδο δηλαδή, που μπορούν να αποκομίζουν. Very much, Mr. Jefferson. Yes. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νότζεμ, ο κύριος Γέπισεν να απαντήσω σε ό,τι αφορά τα Εθνικά Κοινοβούλια και τις έρευνες. Χαίρομαι πάντως που ακούω ότι υπάρχει αυτή η τάση και γίνεται προσπάθεια και στις ε, ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε. Νομίζω ότι μπορώ να σας πω ότι αυτή η προσπάθεια, αυτή η προσοχή ε, φαίνεται ότι δεν έχει καταγραφεί πάρα πολύ στην Ουάσιγκτον, ούτε είναι ε, τα φώτα των προβολέων στραμμένα πάνω σε αυτές τις προσπάθειες. Mm υπάρχει ασύμετρη πληροφόρηση. Είναι πολύ δύσκολο κανείς να επισέλθει στην ουσία, στον πυρήνα του θέματος. Αλλά θεωρώ ότι εμείς ως κοινωνία των πολιτών και ως Ευρωπαίοι πολιτικοί, εσείς, γενικώ εμείς θα πρέπει να το στηρίξουμε αυτό εφόσον μπορούμε. Δηλαδή, να γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε εθνικό επίπεδο γιατί Εκεί ε, λαμβάνονται οι αποφάσεις ε, για τα εθνικά προγράμματα ασφαλείας και εκεί εφαρμόζονται. Το ερώτημα του κυρίου Άλμπερεχτ για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Πάρα πολύ καλά τα είπατε και πολύ σωστά καταλάβατε. Σίγουρα δεν ε, καθησυχάζονται οι Ευρωπαίοι πολίτες σε ό,τι αφορά τους νόμους, τις πρακτικές που με βάση τις οποίες λειτουργούν οι υπηρεσίες οι μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ε, όλα αυτά ε, κρύβονται από ένα πίπλο, πέπλο μυστηρίου. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή διαδικασία και οι κυβερνήσεις ε, θα πρέπει να προσπαθήσουν να εντοπίσουν και να συμφωνήσουν μια δέσμη προτύπων για το πώς τα ευρωπαϊκά προγράμματα πληροφοριών θα σέβονται τις αρχές της σύμβασης. Σίγουρα είναι μακρύς και δύσκολος ο δρόμος προς κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε κανείς ε, να επιβάλλει στις κυβερνήσεις να προχωρήσουν σε ένα τέτοιο μονοπάτι. Το ερώτημα του κύριου Κέρκοπ για την τεχνολογία, την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πράγματι, πολύ ευφύς και εύστοχη παρατήρηση ότι η διαδικασία είναι σταδιακή, εξελικτική. Αυτό που βλέπουμε με τις αποκαλύψεις περί NSA, αυτό που είδαμε είναι τι γίνεται όταν ο νόμος, ε, η πολιτική και η δικαστική εποπτεία δεν καταφέρνουν να παρακολουθήσουν ε, αυτή τη διαδικασία, μένουν πίσω. Πρέπει να βρούμε βέβαια λύσεις. Και μια λύση είναι να υπάρχει επικαιροποίηση των ελέγχων που θα πρέπει να γίνονται στο πλαίσιο των συστημάτων, κάτι που δεν συμβαίνει. Τέλος, τα περί προεπολισμού, νομίζω τα απάντησε ο Γκρέγκ, δηλαδή τα οικονομική τις οικονομικές πτυχές των επιχείρησεων της NSA, νομίζω έτσι, ναι. Ναι, θα ήταν ενδιαφέρον να έχουμε μια ναι, κυρία Ένστη, το ερώτημα της κυρίας Ένστ χωρίς μικρόφωνο βέβαια. Ναι, ναι, συγγνώμη. Νομίζω τα είχα καλύψει για αυτά. Μιλούσατε για τους ελέγχους και τις διασφαλίσεις. Ό,τι έδειξαν οι αποκαλύψεις για την NSA στις ΗΠΑ είναι έλλειψη ελέγχου, έλλειψη εποπτείας, έλλειψη δικαστικού ελέγχου αυτό δείχνουν οι αποκαλύψεις για την NSA ότι και το Αμερικάνικο Κογκρέσο δεν έχει τηρηθεί ενήμερο και το δικαστήριο της ΦΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να έχει το είδος εποπτείας που θα έπρεπε να έχει από την ευρωπαϊκή πλευρά πάλι δεν ξέρουμε αν η κατάσταση είναι καλύτερη ή χειρότερη. Δεν ξέρω αν κανείς έχει τέτοιου είδους πληροφορίες αυτή τη στιγμή ερευνάμε αυτά τα θέματα, αλλά προς το παρόν είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ένα πράγμα θέλω να τονίσω. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των πόρων και των ικανοτήτων που βρίσκονται που υπάρχουν στις Ευρωπαϊκές Υπηρεσίες Πληροφοριών έναντι των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν μια μοναδική θέση και γι' αυτό έχουν και μια μοναδική ευθύνη για όλα αυτά. Πάμε στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Κάποιος θέλει να μιλήσει από την Αμερική. Ναι, συγγνώμη δεν σας άκουσα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Υπάρχει μια έντονη πεποίθηση μεταξύ των μελών της κοινωνίας των πολιτών στις ΗΠΑ ότι αυτοί οι μηχανισμοί που έχουν θεσπιστεί για την εποπτεία της ε, συλλογής πληροφοριών και για την λογοδοσία των υπευθύνων έχουν αστοχήσει, έχουν αποτύχει και παρόλα αυτά ήταν πολύ στεναροί και ισχυροί μηχανισμοί. Αγωνιζόμαστε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Γιατί αυτοί οι μηχανισμοί έγιναν ακριβώς για να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπήρχε υπερβολική παρακολούθηση που να περιλαμβάνει και παρακολούθηση για τα πολιτικά φρονήματα. Το γνωρίζανε αυτό όμως και δεν το αποκαλύψανε τότε οι υπηρεσίες πληροφοριών. Όλοι περιμέναν ότι αργά ή γρήγορα θα βγουν στη φόρα όλα αυτά τα πράγματα. <clears throat> Όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν επικριτές του προγράμματος του τίτλου 215 προβλέπαν ότι κάπου θα βγουν στη φόρα όλα αυτά και θα υπήρχε μεγάλο σοκ στην κοινωνία. Αυτό έγινε. Σε κάποια στιγμή η Επιτροπή για τις Υπηρεσίες Πληροφοριών στο Κογκρέσο δεν έδωσε τον φάκελο στους απλούς βουλευτές του, του Κογκρέσου, ώστε να μην ξέρουν για τις δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών που θα εγκρίνανε και πάλι. Αυτό ήταν μεγάλη αστοχή από τη δική τους πλευρά. Και το δικαστήριο της Φάιζα, το οποίο θα πρέπει να εγκρίνει την εποπτεία αυτή, πολλές φορές ήταν στο σκοτάδι και δεν ήξερε ακριβώς τι είδους διαδικασίες <clears throat> παρακολούθησης λαμβάναν χώρα. Η κυβέρνηση και η NSA πηγαίνουν στο δικαστήριο αυτό και λέγανε ότι εμείς ψάχνουμε να βρούμε μονάχα το ιστορικό των τηλεφωνικών ε, συνδιαλέξεων μόνο όταν πετύχουμε ένα επίπεδο που είναι αρκετό για να προστατεύσει την ιδιωτικότητα. Αλλά φάνηκε με τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι αυτό ήταν μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας να κάνουν προσπάθειες να προστατεύσουν τις ε, ιδιωτικές Υπάρχει λοιπόν παράκαμψη του, της εποπτείας των δικαστηρίων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο μόνος τρόπος να γίνει κάτι για όλα αυτά είναι να υπάρξει ε, περιορισμός της ε, συλλογής πληροφοριών από τον νόμο και να μην επιτρέπεται η χίδιν συλλογή στοιχείων όπως γίνεται τώρα. Um... Ευχαριστώ πολύ. Ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο γύρο ερωτήσεων. Καθυστέρησαμε λιγάκι. Σας παρακαλώ να είσαστε λίγο συντομότεροι δύο λεπτά το μέγιστο. Αν μπορείτε να είστε πιο σύντομοι, ακόμα καλύτερον. Ζίπελ, Γκόμες, Βαϊνάχτες και Μπρόντς. Κάποιος άλλος? Η κυρία Μορβάη. Κλείνω. Κυρία Ζίπελ. Προσπαθώ να είμαι σύντομη. Κύριε Γέπεσε, νομίζω στις απαντήσεις σας είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Όταν λέτε ότι πρέπει να προσαρμόσουμε πάντα τους μηχανισμούς ελέγχου και εποπτείας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχει παραμεληθεί στο παρελθόν, ιδίως μετά τα γεγονότα της 11 η Σεπτεμβρίου και αν δούμε την έκταση της παρακολούθησης που γίνεται, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι τα εμπορικά συμφέροντα βρίσκονται στο κέντρο της ε, αντιμετώπισης και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με δημόσιες ελευθερίες και η ιδιωτική ζωή έχει σπροχτεί στο περιθώριο. Εσείς είπατε τώρα ότι στην αρχή αρχίζει να υπάρχει μια αντίσταση στο νόμο, στην νομοθεσία Patriot και στο νόμο για τη ΦΙΖΑ σε ό,τι αφορά τα νομικά θέματα, όμως θα πρέπει ακόμα και οι νόμοι για την εποπτεία να επανεξεταστούν και κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει κάποια ελπίδα να υπάρξει αυτή η αλλαγή της νομοθεσίας στις ΗΠΑ και η προσαρμογή της στην προστασία των δικαιωμάτων. Κυρία Ευχαριστώ πολύ. Στο Twitter διαβάζω ότι η Τίλμα Ρουσέφ από τη Βραζιλία μιλάει ε, ε, πριν από τον Ομπάμα, που μίλησα μάλλον πριν από τον Ομπάμα στην ε, Γενική Συνέλευση του είπε ότι δεν είναι μόνο η παρακολούθηση παράνομη, αλλά παραβιάζει κατάφορα και το διεθνές δίκαιο, τους διεθνούς κανόνες και την κυριαρχία ακόμη, την εθνική. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω το εξή ερώτημα. Αν πράγματι υπήρξε αυτή η αποτυχία, δεν υπήρξε δηλαδή έλεγχος, δεν υπήρξε εποπτεία ε, στο Κογκρέσο. Αυτό δεν συνέβη γιατί δεν υπήρχε μηχανισμός, όπως είπαν οι ομιλητές μας, Τζέπισεν και Νότζιμ. Αυτά συνέβησαν γιατί υπήρξε πρόβλημα κεραιότητας, ήταν θέμα πολιτικής ε, αφέλειας, μακιαβελισμός, ε, κινησμός, τι ήταν. γιατί οι επιτροπές πληροφοριών, τα intelligence committees, γι' αυτό το λόγο συγκροτούνται και απέτυχαν. Πώς λοιπόν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο θα έχουμε ένα παρόμοιο σύστημα που δεν έχουμε. Κάποια εθνικά κοινοβούλια ίσως ναι, αλλά τα περισσότερα εθνικά κοινοβούλια δεν έχουν κάτι αντίστοιχο και δεν λειτουργεί. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουν ε, αυτό που έχουν αναλάβει να κάνουν. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και πράγματι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα ιδιαίτερο ρόλο στα θέματα αυτά. Λίγα κοινοβούλια έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τόσο έντονα όλη αυτή την προβληματική. Τώρα, αυτό το οποίο αναφέρατε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας γενικός διατλαντικός διάλογος πέραν όλων των άλλων πολιτικών θεμάτων. Υπάρχει το θέμα της ε, τεχνολογικής εξέλιξης που θα πρέπει κάπου να ελεγχθεί πέρα από τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Θα ήθελα να ξέρω πώς βλέπετε αυτό το διατλαντικό διάλογο, με ποιους εμπλεκομένους, με ποια ζητήματα συζήτησης και ποιο ρόλο θα πρέπει να έχουν και οι συζητήσεις στην Ευρώπη για το πακέτο για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων που τώρα εμείς <clears throat> θα εγκρίνουμε. Bronze. Ναι. Η συλλογή δεδομένων, ιδίω προσωπικών δεδομένων, είναι πάντα μια εισβολή στην ιδιωτική ζωή. Εγώ έχω λιγότερα μυστικά από ό,τι είχα παλιότερα, αλλά όλοι μας νιώθουμε αυτήν την εισβολή όταν χρησιμοποιούνται αυτά τα δεδομένα για τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Η χρήση των δεδομένων είναι ένα πολύ πιο σημαντικό θέμα από το θέμα της συλλογής τους. Πριν από δύο-τρεις εβδομάδες Ρώτησα τον κύριο Applebaum αν οι πληροφορίες οι οποίες έχουν συλλεχθεί χρησιμοποιήθηκαν για καθαρά πολιτικές αντιπαραθέσεις και μεταξύ κρατών μελών και μέσα σε κράτη-μέλη. Και που είπε ότι το πρόγραμμα αυτό συλλογής πληροφοριών ασχολείται περισσότερο με πολιτικές διαμάχες και πολιτικά προβλήματα και σκασίλα του περίπου η τρομοκρατία και λέει ότι με αυτόν τον τρόπο παίζουν και κάποιο ρόλο στο να νομιμοποιούν διεθνείς επιθέσεις. Και ίσως πρέπει να προσθέσουμε μία ακόμα αίτηση σε αυτά που είπε ο κ. Τζέφεσον, ότι οι πληροφορίες οι οποίες συλλέγονται δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να επηρεάσουν την κοινή γνώμη σε εκλογικές εξαρτίες σε χώρες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την τρομοκρατία. Ευχαριστώ. Κυρία Μορβάη, τελευταία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να προσεγγίσω αυτό το θέμα κάπως διαφορετικά. Να αναδιατυπώσω την ερώτηση του κ. Μπρόνζ. Σύμφωνα με τους προσκεκλημένους μας όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν συλλεγεί παράνομα, για ποιο λόγο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία των Ευρωπαίων πολιτών, τι τα κάνουν. Έπειτα, άλλη ερώτηση. Υπόθηκε ότι τελικά δεν κερδίζουν και πολλά χρήματα αυτές οι εταιρείε που εμπλέκονται σε αυτή την... είναι ας πούμε υπεργολάβη της Αμερικανικής Υπηρεσίας ε, Πληροφοριών. Πώς είναι δυνατόν, γιατί δεν μπορώ να τώρα να σας δώσω ακριβώς την παραπομπή, αλλά θα μπορούσα, πώς γίνεται να δημοσιεύεται το γεγονός ότι τα μέλη του Κογκρέσου και ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουν δεν σχετίζεται με το κατά πόσο ανήκουν σε συγκεκριμένες ε, ομάδες, αλλά από τα ποσά που έχουν λάβει για τις εκστρατείες. Και μάλιστα ποσά που έχουν λάβει από αυτές τις ίδιες τις επιχειρήσεις που κάνουν την ε, υπεργολαβία. Δεν, μας, δεν πρέπει να μας ε, περνάνε και για ηλίθιους. Ο, μόνο χάρη στον Έντουαρ Σόντερ να έχουμε αυτές τις πληροφορίες. Πώς μπορεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να προστατεύσει την ασφαλεία της στο μέλλον. Ναι. Να σας ζητήσω να απαντήσετε σε αυτά τα ερωτήματα. Και επειδή τελειώνει ο χρόνος μας, παρακαλώ να είστε σύντομοι, γιατί έχουμε άλλη συνεδρία και άλλη ε, βιντεοδιάσκεψη. Θέλεις να μιλήσεις πρώτα για τα σημεία που αφορούν τη ΣΥΠΑ? Όχι, όχι, μετά από σένα. εμπορικά συμφέροντα. Από όσα γνωρίζουμε, δεν φαίνεται να υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα άμεσα πίσω από τις δραστηριότητες της NSA. Αλλά είναι πολύ πιθανό ένα από τους τρόπους ε, αντιμετώπισης της, των δραστηριοτήτων της NSA να είναι μέσω εμπορικού αντίκτυπου. Οι εταιρείε ίντερνετ και cloud ήδη αισθάνονται την απώλεια της εμπιστοσύνης των καταναλωτών παγκοσμίω. Τώρα, για τον Ιατλαντικό, περατλαντικό διάλογο και την, το κατά πόσο οι κυβερνήσεις μπορούν να βρεθούν σε μία αίθουσα και να συζητήσουν, είναι καλό το ερώτημα, αλλά δεν έχουμε απάντηση για το πώς θα τις δώσουμε τα κίνητρα ή θα τις παροτρύνουμε να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Κογκρέσο και Κοινοβούλιο. Αυτή η συζήτηση γίνεται νομίζω. Υπάρχουν ανταλλαγές. Right. Well, we can only, I mean, we can only encourage that, that sort of a debate. Mr. Bruns raised, and, and, and the last speaker as well, raised the question about collection. Τελευταίος ομιλητής μίλησε για τη συλλογή και χρήση των ε, στοιχείων αυτών. Αυτό που βλέπουμε εν γέννη, καθώς βλέπουμε αυτά τα προγράμματα παρακολούθησης, είναι ε, να, ότι μειούται η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους χρήστες ε, που χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυστηρά για την εθνική ασφάλεια και τις άλλες χρήσεις. Νομίζω αυτά έχω να πω. Να δούμε αν ο Γκρέγκ έχει άλλα σχόλια. Ευχαριστώ. Κύριε Νόιζιν, έχω δύο πράγματα να πω. Οι κατευθύνσει γραμμέ ελαχιστοποίηση που διέπουν την παρακολούθηση σύμφωνα με το πρόγραμμα Πρίσμα δεν μπορούν ε, και επιτρέπουν ε, να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία αυτά για οποιοδήποτε νόμιμο σκοπό. Δηλαδή, εάν δεν απαγορεύεται συγκεκριμένα ρητά με τον νόμο, η χρήση του ε, επιτρέπεται. Αυτό είναι πολύ ευρύ, αλλά δεν έχω ακούσει να γίνεται καμιά προσπάθεια στο Κογκρέσο για να προσθεθεί κάποια νέο περιορισμό για τη χρήση αυτών των πληροφοριών. Εμείς συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει οικονομικό κίνητρο ώστε οι εταιρείε να κάνουν παρακολούθηση, να πληρώνονται εντάξει για την, όταν υποχρεούνται να το κάνουν, αλλά δεν θα πρέπει να είναι τεράστια η αμοιβή γιατί φυσικά αυτό δημιουργεί κίνητρο που είναι αντίθετο προς την ίδια τη δομή που έχει στόχο να προστατεύει τον ιδιωτικό, την ιδιωτικότητα. Δηλαδή ότι η εταιρεία κάνει μόνο την ε, παρακολούθηση που τη ζητά η κυβέρνηση. Ε, νομίζω λοιπόν πως θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες πληροφορίες για όλα αυτά και προσπάθειες ε, στο Αμερικανικό Κογκρέσο ώστε να εξασφαλιστεί ότι μόνο το κόστος τους θα καλύπτεται. Δεν θα δημιουργείται δηλαδή κάποιο οικονομικό όφελος ώστε να θέλει κανείς να κάνει αυτή τη δουλειά της παρακολούθησης. Τώρα, διαφάνεια λύπη. Λύπη, γιατί γι' αυτό έχουν δημιουργηθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Ας πούμε το, το δικαστήριο Φάιζαντ έδωσε κάποιες ονομοδοτήσεις, αλλά όσον αφορά τη συμπεριφορά των εθνικών υπηρεσιών ασφαλείας. Μα σε ποιους τα έστειλαν όμως αυτά. Ε, τα στείλαν στους ίδιους που κάναν την παρακολούθηση, εναντίον των οποίων αποφάσισε και γνωμοδότησε το ίδιο το δικαστήριο. Έχουμε κάποιες ελπίδες, ιδιαίτερα για την έννοια ότι οι γνωμοδοτήσεις αυτού του δικαστήριου θα πρέπει να δημοσιεύονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γέπισεν και κύριε Νόζιμε που ήσασταν μαζί μας από την άλλη όχθη του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ όλους. Τελειώνει έτσι η τρίτη συνεδρία και περνάμε στην τέταρτη. Αποτελεσματικότητα της παρακολούθησης, τα πολέμηση του εγκλήματος και ε, της τρομοκρατίας στην Ευρώπη. Περιμένουμε μια άλλη τηλεδιάσκεψη, δεν ξέρω αν είναι στα έτοιμη. Δύο λεπτά. In time I I'll explain ε, whom we'll be listening to. Mr. Reinhard Kreisel from Θα ακούσουμε τον κύριο Κράισλερ, που είναι συντονιστής του προγράμματος IRIS. And IRIS means increasing resilience. Άρη σημαίνει αυξανόμενη ανθεκτικότητα στις κοινωνίες ε, παρακολούθησης. Και μετά από την παρουσίαση θα έχουμε μια περίοδο ερωταπαντήσεων. Κύριε Γκράισερα, μπορούμε να σας δούμε. Καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας ακούτε? Εμείς δεν ακούμε πολύ καλά πάντως. So welcome to the session of the LIBE Committee in the European Parliament. I um, will immediately give you the floor because we've kept you waiting uh, for a bit. Σας ακούμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα παρακολουθήσουμε πρώτα την παρουσίασή σας και στη συνέχεια θα σας θέσουμε ερωτήματα και θα έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε. Έχετε το λόγο για την παρέμβαση σας. Μπορούμε να μιλήσουμε για τα θέματα της παρακολούθησης σε δημοκρατικές κοινωνίες. Δεν υπάρχει πολύς ε, χρόνος, βέβαια. Η εποπτεία για την παρακολούθηση τώρα του εγκλήματος Δυστυχώς ο ήχος δεν είναι πολύ καλός και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέει ο μιλητής, αλλά δεν είναι ο κατάλληλος ήχος για τέτοιου είδους ε, συνεδρίες. Ε, υπάρχουν τα λεγόμενα μηχανικά αναγνώσιμα κοινωνικό ε, τεχνικά υβρίδια τα οποία αντιμετωπίζουμε. Οι εταιρείε αυτές λοιπόν για την παρακολούθηση χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων. αν χρησιμοποιούνται τώρα αυτές οι τεχνολογίες για να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία. Αυτές οι τεχνολογίες είναι χαμηλού επίπεδου, μπορούν να αντιμετωπίσουν άτομα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επίσης για, για άλλους στόχους και μεταξύ των οποίων...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 κατά ένα-δύο λεπτά. Σας παρακαλώ λοιπόν να ολοκληρώσετε εδώ και επειδή έχει ζητήσει ήδη ερώτημα να θέσει ο Κλοντ ή μάλλον είπε ότι δεν θα θέσει ερώτημα τελικά και για να μείνουμε στο χρόνο έχω τους δύο σκιώδες μπροστά μου θέλω να τους πω θέλετε το λόγο εσείς και ποιος άλλος θέλει το λόγο δύο έχω ήδη Κύριε Φως, θέλετε να κάνετε ερώτημα ο σκιώδης. Sorry. ich hatte auf Deutsch oder Englisch? Γερμανικά ή αγγλικά. Yeah. Ε, um... Ε, Καταλαβαίνω γερμανικά λέει και ο προσκεκλημένος. Είχα δύο ερωτήματα. Δύο ερωτήματα σε ένα. Η παρακολούθηση αυτή συνίσταται κατά την ειδική σας άποψη και σε παρακολούθηση ιδιωτικών εταιριών που αναλύεται η συμπεριφορά τους λεπτομεριακά. Το δεύτερο ερώτημα, μήπως έχετε την εντύπωση ότι ούτως ή άλλως ζούμε σε ένα κόσμο με όλο και μεγαλύτερο επίπεδο παρακολούθησης, γιατί με τη τεχνολογική ανάπτυξη υπάρχει όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα παρακολούθησης ιδιωτικής ζωής. Κυρία Ένστ επίσης. Και μετά η κυρία Ζίπελ και ο κύριος Μπρόνς θέλουν το λόγο. Σας ζητώ να κλείσουμε τον κατάλογο ομιλητών. Κυρία Ένστ. Και εγώ πάρα πολύ σύντομα. Πώς μπορεί κανείς να αλλάξει τη λογική ώστε να περάσουμε από αυτή την κοινωνία της παρακολούθησης, να αποσυνδεθούμε από αυτή τη λογική της συνεχούς παρακολούθησης και αστυνόμευσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι μαζικών παραβιάσεων. Και το δεύτερο είναι αυτό που έχει να κάνει με τους μηχανισμούς ελέγχου σε σχέση με την εποπτεία αυτή. Μπορείτε να πείτε κάτι για τις δυνατότητε που πιστεύετε ότι μπορούν να γίνουν σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι έχει αποτύχει μέχρι στιγμή, αλλά για το μέλλον τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, κυρία Ζήπελ. Μόνο ένα ερώτημα, θέλω να θέσω. Μιλήσατε για το κίνδυνο ότι οι ανοιχτέ συζητήσει δεν θα είναι πια δυνατέ γιατί όλα παρακολουθούνται και όλα καταγράφονται. Το μόνο μου ερώτημα είναι το εξή. Θα επηρεάσει αυτό και την τελείως ιδιωτική ζωή των ατόμων. Γιατί κάθε φορά που γίνω στο ίντερνετ σε ένα, κοινωνικό δίκτυο πιστεύετε ότι ακόμα και οι πιο ιδιωτικές ε, στιγμές θα παρακολουθούνται και θα αναγκαστεί ο κόσμος να αλλάξει τη συμπεριφορά του όταν έχουμε μια τόσο μαζική παρακολούθηση μπρόνς. Μάλιστα. Ποιο είναι το ποσοστό των σχεδιαζομένων τρομοκρατικών ενεργειών που έχουν αποτραπεί από τις ενέργειες παρακολούθησης έναντι αυτών που ήταν επιτυχείς ή που απέτυχαν επειδή ήταν ασχετικές κιτζίδες οι τρομοκράτες ή επειδή τα πράγματα απλώς δεν δούλεψαν σωστά. Είχα και εγώ να θέσω ένα ερώτημα. Αν καταγράψετε την αποτελεσματικότητα οποιοδήποτε. Σε αυτήν την περίπτωση την αποτελεσματικότητα της εποπτείας. Μπορείτε να το κάνετε μονάχα αν συγκρίνετε το αποτέλεσμα έναντι του προσδοκούμενου αποτελέσματος και του κόστους. Άμα δεν ξέρετε όμως τι προσδοκείτε, πώς μπορείτε να πείτε ότι είναι αποτελεσματική και άμα δεν ξέρετε ποιο είναι το κόστος. Και όταν υποτίθεται ότι αυτή η παρακολούθηση είναι για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και δεν μας λένε τίποτα οι υπηρεσίε πληροφοριών για τις επιθέσεις οι οποίες έχουν αποτραπεί. Πώς μπορούμε να έχουμε οποιαδήποτε αξιόπιστη αξιολόγηση σε σχέση με την αποτελεσματικότητα ή ου αυτής της παρακολούθησης. Έχετε λοιπόν πέντε ερωτήματα, εάν θα μπορούσατε να απαντήσετε όλα μαζί και θα κλείσουμε. Let me start from the end. This is precisely the problem, say, how to measure prevention, how to measure a non-event, to measure a non-event. And this is a debate that's been going on among law enforcement and their critics for quite some time.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 vocabulary or conceptual background to really understand this. Um, can, the logic... can, I, can I ask you to wind up a little bit as we have the... Μπορείτε να συντομείτε σας παρακαλώ να ολοκληρώνετε γιατί έχουμε και έναν ακόμη γύρο, μια ακόμα συνεδρία. Συγγνώμη, αλλά πρέπει να έχω υπόψη και την ώρα. What can be done to change the logic uh, in parliamentary terms? Uh, Good question. I think we had this this infamous INDEC project that was scandalized by the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 κατανοώ ότι όταν, δεν έχει, όταν έχει μια βιντεοσύνδεση δεν μπορεί διακριτικά να κάνει ένα ανέβημα στον ομιλητή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και για την παρουσίασή σας και την απάντηση, τις απαντήσεις που δώσατε στα ερωτήματά μας. Ερχόμαστε λοιπόν στην τελευταία συνεδρία, συνεδρία υπαριθμών 5, με τον κύριο Κάσπαρ Μπάλτεν, που είναι γνωστό σε πολλούς από εσά από προηγούμενες ε, ακροάσεις επιτροπής μας ο κύριος Μπάλτεν έχει προετοιμάσει και μία μελέτη για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα τη δείτε στα γραφεία σας, στα έδρανά σας. Προγράμματα παρακολούθησης των ΗΠΑ και επίπτωση στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας κάνει μία σύντομη εισαγωγή. Μακρά εισαγωγή. Όχι καμία εισαγωγή λέει ο κύριος Μπάλτεν. Δεν πρόκειται να, δεν πρόκειται να κάνω καμία εισαγωγή. Εντάξει. Για αυτούς οποίους, οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το, την έκθεση του κύριου Μπάλτεν και άλλων, για τους ελάχιστους που δεν την έχουν διαβάσει, ίσως μπορείτε να τους δώσετε μια πάρα πολύ μικρή και κούτσικη εισαγωγή, δύο-τρία λεφτά που να περιέχει τα κύρια συμπεράσματα. όλοι από εμά ξέρουμε τη θεματολογία, αλλά όχι όλοι. Και μετά αρχίζουμε τη συζήτηση με την άδειά σας. Πήρα μια διαφορετική προσέγγιση. Είχα κάνει μια παρουσίαση το Φεβρουάριο για αυτή την έκθεση. Αυτή η έκθεση έχει σαν στόχο να είναι συνοπτική και <clears throat> να είναι ε, αυτάρκης και να στέκεται μόνη της. Να κάνουμε μια πιο διαφορετική προσέγγιση αν θέλετε, να εστιάσουμε στα θέματα τα οποία ενδιαφέρουν περισσότερο την Επιτροπή σας υπάρχουν μερικά πολύ σημαντικά στοιχεία που βρίσκονται μέσα στην έκθεση και θα ήταν για μένα πιο παραγωγικό να σταθούμε σε αυτά συγκεκριμένα σημεία. Μπορεί κάτι να χαθεί, αλλά θα ήταν πιο αποτελεσματικό και η χρήση του χρόνου παρά να προσπαθώ να σας πω και πάλι αυτά τα οποία θα βρείτε ούτως ή άλλως. Εντάξει, δικό σας είναι ο λόγος και μπορείτε να αποφασίσετε ό,τι θέλετε. 15 λεπτά και μετά πάμε ερωτήσεις και απαντήσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνει το κοινοβούλιο, μου το κοινοβούλιο και η επιτροπή σα να ετοιμάσω αυτή την έκθεση. Η έκθεση αυτή αφορά μονάχα τι δραστηριότητε των ΗΠΑ και τη Εθνική Υπηρεσία Ασφάλεια NSA των ΗΠΑ. Φυσικά υπάρχει σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων των ΗΠΑ και τη NSA και των δράσεων κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό δεν ήταν αντικείμενο τη έκθεση. Δεύτερον, εγώ θεωρούμε ότι είμαι πάντα ο κύριος σύμβουλος ασφαλείας της Microsoft για να μην υπάρχουν παρεξήγησεις. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ των δικών μου απόψεων και των απόψεων της Microsoft, αν έχετε αυτή την εντύπωση. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω έχει γενικότερο χαρακτήρα και απευθύνεται σε κάτι που είπε ο κύριος Μπρόντς προηγουμένως μπορεί να, νομίζουν ότι η συλλογή δεδομένων είναι λιγότερο σημαντική από τη χρήση των πληροφοριών. Εγώ διαφωνώ. Και γιατί διαφωνώ. Μετά από τις αποκαλύψεις του Edward Snowden, η κοινή γνώμη τώρα κατανοεί ότι κάποια άτομα που έχουν υψηλή θέση στην κοινωνία, πολιτικοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες, γνωρίζουν ότι η NSA κατά πάσα πιθανότητα γνωρίζει όλα τα προσωπικά τους ε, μυστικά, εάν έχουν περάσει σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο. Δεν ξέρουμε πόσα χρόνια πίσω μπορεί να κρατήσει αυτό το θέμα. Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ αποσταθεροποιητική κατάσταση στις δημοκρατίες μας. Γιατί αυτό σημαίνει ότι η κοινή γνώμη θα πρέπει να σκεφτεί αν αυτά τα άτομα κοιτάνε πίσω από τον νόμο τους και λένε μήπως δεν πρέπει να το πω αυτό, μήπως θα πρέπει να τα πω λίγο πιο ήπια, μήπως δεν θα πρέπει να κάνω κάτι το οποίο θα προσκρούσει στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Γιατί αν έχουν αυτοί οι άνθρωποι μυστικά τα οποία είναι γνωστά στην NSA, είναι κατά κάποιο τρόπο εκδιάσιμη. Αν πιστεύει κοινή γνώμη ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα να είναι εκδιάσιμη, αυτό είναι κάτι το οποίο ήδη έχει μια μεγάλη σημασία και αυτό είναι μια αλλαγή η οποία έχει γίνει και δεν το έχουμε ακόμα συνειδητοποιήσει απόλυτα λόγω της έκτασης των αποκαλύψεων Σνόντεν. <clears throat> Ένα δεύτερο σχόλιο. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα δεκάδες χιλιάδες εγγράφων από τις αποκαλύψεις του κ. Σνόντεν που δεν έχουν παρουσιαστεί και δεν έχουν αναλυθεί. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό ότι όλα αυτά τα στοιχεία που βρίσκονται στην έκθεσή μας δεν είναι τίποτα, είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στις αποκαλύψεις που μπορεί να ακολουθήσουν. Εμείς προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε πληροφορίες ιστορικού χαρακτήρα και το γενικό πλαίσιο για να τα συνδυάσουμε με τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει το, τα, τελευταίους μήνες. Στη σελίδα 8 το πρώτο ζήτημα που θέλω να φέρω στην προσοχή σας είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολλές φορές το ξεχνάμε. Η διακυβέρνηση της ιδιωτικής προστασίας το πώς λειτουργεί η νομοθεσία προσωπικών δεδομένων. Αν το δείτε ιστορικά, γίνεται κάτι παράξενο για αυτό την νομοθεσία, γιατί αφαιρεί κάτι το οποίο είναι μια ουσιαστική εξουσία από τους πολίτες. Μόλις οι πληροφορίες πάνε σε ένα άλλο σύστημα, είτε είναι ένα σύστημα στον ιδιωτικό τομέα, είτε σε κυβερνητικό, κυβερνητική δάση δεδομένων, δεν μπορεί να έχει καμιά αντίρρηση ο πολίτης αν θα μεταγραφεί και θα αντιγραφεί για χίλιους διαφορετικούς, σε άλλες χίλιες διαφορετικές βάσεις δεδομένων, σε άλλες χώρες, σε άλλες εταιρείε που έχουν ένα διαφορετικό νομικό καθεστώς. Λοιπόν, εάν έχει γίνει η απαραίτητη νομική διαδικασία σε τυπικό επίπεδο, ο πολίτης δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αλλά ξέρουμε ότι κάθε φορά που μεταγράφεται αυτή η πληροφορία αυξάνει, αυξάνει μονοτονικά ο κίνδυνος, δεν μειώνεται ποτέ είναι πολύ πιο πιθανό να γίνει κάτι με τα δεδομένα και επομένω κάτι μπορεί να γίνει με το άτομο που αφορούν τα δεδομένα. Εδώ και πολλά χρόνια στην προστασία δεδομένων αυτό θεωρείται δεδομένο. Αλλά με τις ε, αποκαλύψεις Snowden και με τη χρήση του υπολογιστικού νέφους ίσως πρέπει να θέσουμε και περαιτέρω ερωτήματα σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων και την νομοθεσία. Κοιτάζοντας την έκθεση, έρχομαι στη σελίδα 13 στο, για το XKey, το οποίο είναι ένα σύστημα ταξινόμησης που έχει στοιχεία τριών ημερών που αλλάζουν κάθε, που ενανεώνονται σε 150 παγκόσμια κέντρα. Έχει ε, διευθύνσεις email, έχει ονόματα ε, ανθρώπων, έχει διευθύνσεις IP κτλ αυτός ο δείκτης. Αυτή είναι μια παρουσίαση που δεν σας φαίνεται να σημαίνει τίποτα, αλλά καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι η ικανότητα παρακολούθηση που μπορεί να προκύψει από το σύστημα αυτό του 6 είναι κάτι το οποίο εμεί δεν μπορούμε να το συλλάβουμε και ο Όρουελ δεν μπορούσε να το είχε ανθιστεί ποτέ στη ζωή του. Έχει λοιπόν αναλυτήσει ένα είδος μηχανή του χρόνου ώστε ακόμα και δεν έχει καμία υποψία για ένα άτομο, μπορεί να γυρίσει πίσω και να αναλύσει όλη τη ζωή, όλη την ε, ε, πολιτεία αυτού του ανθρώπου από την αρχή της ζωής του. Βέβαια αυτό δεν αφορά τους Αμερικανούς. Στη σελίδα 14 το πρόγραμμα ε, που χρησιμοποιεί η NSA για να σπάει συστήματα κρυπτογράφησης, όχι κατευθείαν βέβαια, αλλά ε, με μαθηματικές τεχνικές χρησιμοποιώντας ε, τις ε, ηλεκτρονικές, το ηλεκτρονικό θόρυβο από τον υπολογιστή από όπου μπορεί να βρει το κλειδί και επίσης με το να διαφθείρει τη, τα προγράμματα των εταιριών λογισμικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει δημιουργήσει μεγάλο σοκ σε παγκόσμιο επίπεδο και προσπαθούν τώρα να δουν οι ειδικοί τη πληροφορική ποια συστήματα μπορεί να είναι τροτά σε τέτοιου είδου επιθέσει. Αλλά δουλεύουν ακόμα στο σκοτάδι. μιλώντα με κάποιου δημοσιογράφου που είχαν πρόσβαση σε αυτό το υλικό, εγώ προσωπικά δεν είχα, δεν μπορούμε να περιμένουμε να βγουν πιο λεπτομεριακά στοιχεία. Έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Ξέρουμε ότι πολλά από τα συστήματα που θεωρούσαμε πριν από τρει μήνε ότι ήταν ασφαλή, τώρα ξέρουμε ότι ένα μεγάλο μέρο από αυτά είναι επισφαλή. Αλλά δεν ξέρουμε ποια είναι αυτά που είναι επισφαλή. Συνεχίζω. Στη <clears throat> σελίδα 18, πληροφορίες ε, τύπου Foreign Intelligence, δηλαδή πληροφορίες που αφορούν ξένες χώρες. Αυτά ξεκίνησαν με το νόμο του 1978 για τις πληροφορίες από, από τρίτες χώρες και το βασικό στοιχείο αυτού του νόμου δεν έχει αλλάξει από το 1978. χρειάζεται να αλλάξετε δύο επίπεδα ορισμών σε αυτά που έχετε εδώ. Και μόνο το ένα δέκα, δέκατο της ε, πληροφορίας καλύπτουν αυτά. Η foreign intelligence είναι πληροφορίες σε σχέση με ένα πολιτικό φορέα που βρίσκεται στο εξωτερικό ή για ξένο έδαφος που συνδέεται με ή έχει κάποια σχέση ή είναι απαραίτητο για ένα Αμερικανό σε ό,τι αφορά την ε, λειτουργία της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι τεράστια η ευρύτητα αυτού του ορισμού. Σχεδόν όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν κάποια σχέση με την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ ε, περιλαμβάνεται εκεί, ακόμα και η νόμιμη πολιτική δράση των Ευρωπαίων πολιτών. Δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό εφαρμόζεται αυτό στην πράξη, γιατί δεν έχει γραφτεί τίποτα για όλα αυτά εδώ και 40 χρόνια, καμία νομική ερμηνεία, καμία προεδρική διαταγή, καμία ερμηνεία για το τι σημαίνει αυτό. Όλα αυτά δεν ξέρουμε πώς έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 40 χρόνια, αλλά μπορούμε να υποθέσουμε ότι αυτή είναι η βάση με την οποία έχει την εξουσία αυτή η διαδικασία ε, παρακολούθησης είναι ένα είδος πολιτικής κατασκοπίας στα θέματα αυτά. Μέσα σε αυτόν τον ορισμό βλέπετε μία διάκριση επί τη βάση εθνικότητας. Εάν αφορά ένα Αμερικανό πολίτη, θα πρέπει να είναι απαραίτητη αυτή η συλλογή πληροφοριών. Εάν όμως είναι κάτι που δεν αφορά ένα ε, ε Αμερικανό πολίτη, αρκεί να είναι κάτι το οποίο έχει κάποια σχέση με την ε, Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Αν συνδυάσετε τα δύο, υπάρχει μια διπλή διάκριση επί τη βάση της ε, εθνικότητα που δίνει πλεονεκτήματα στου Αμερικανού και μόνο μειονεκτήματα στου άλλου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα αντίστοιχο στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και εδώ δεν έχω μιλήσει καθόλου για ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά μιλώντα για του εμπειρογνώμονε θεωρούν ότι ήδη αυτή η διάκριση είναι παράνομη βάση τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στο 2.1.5, <clears throat> όπω είπε ο Γκρέτ Νόιμαν, Υπάρχουν προσπάθειες για να τροποποιηθεί ο νόμος περί πατριωτισμού, το, η παράγραφος 2.15. Αυτά όμως δεν πρόκειται να μας βοηθήσουν πάρα πολύ, γιατί βλέπετε ένα τμήμα εδώ πέρα το οποίο μάλλον θα παραμείνει ε, ως έχει άθικτο. Υπάρχει πολύ ευρεία ε, άδεια συλλογής ε, πληροφοριών που δεν έχουν να κάνουν με Αμερικανούς πολίτες ε, όταν πρόκειται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ακόμα και αν περιορίσουν λοιπόν την επιλεκτική συλλογή ε, για τους Αμερικανούς πολίτες, αυτό δεν πρόκειται να επηρεάσει καθόλου συλλογή πληροφοριών για τους μη Αμερικανούς πολίτες. Πηγαίνω σε σελίδα 21. Όταν εξετάζουμε <clears throat> τη συλλογή πληροφοριών του τύπου Foreign Intelligence που βασίζεται στο, στο νόμο 702, υπάρχει ο κανονισμό το καταστατικό για όλα αυτά, που λέει πρέπει να υπάρχει μια ελαχιστοποίηση στη στοχοποίηση και τι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται. Όταν τα είχα παρουσιάσει αυτά στη Λίμπε το Φεβρουάριο, δεν περίμενα να δω αυτές τις διαδικασίες, αλλά έχουν τελικά δημοσιευτεί από την Guardian στις 20 Ιουνίου. Όταν διαβάσει αυτές τις διαδικασίες, αυτό που βλέπει είναι ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως περιορισμός και καμιά απολύτως μορφή προστασίας για τους μη Αμερικανούς πολίτες, όπως ειλικρινά το είχα προβλέψει. Αυτό είναι λοιπόν μια πλήρης επιβεβαίωση ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία ή διασφάλιση για τους μη Αμερικανούς. Το άλλο σημείο στη σελίδα 22 έχει να κάνει με μια αποκάλυψη που έγινε στον Αύγουστο 20, 21 Αυγούστου και αυτό ήταν μια επιστολή της Αμερικανικής κυβέρνησης προς τους αρχηγούς της Επιτροπής για τις Υπηρεσίες Ασφαλείας του Αμερικανικού Κογκρέσου. Υπάρχει μια παράγραφος που έχει μεγάλη σημασία για τα θέματα αυτά και η οποία δεν έχει τύχει σχολιασμού αλλού. Τι γίνεται εδώ. Από τη στιγμή που η NSA έχει φιλτράρει τις πληροφορίες που συλλέγει από τα διάφορα συστήματα που αναφέραμε προηγουμένως, εφαρμόζουν ένα σύστημα για να υπολογίσουν με πιθανότητα 50% αν αυτή η πληροφορία αφορά Αμερικανούς. Η πληροφορία που είναι κατά 50% πιθανότητα για τους ξένους συνεχίζει το δρόμο της και την επεξεργασία. Λέει όμως ότι η παράγραφος αυτή μπορεί να σπάσει αυτή η ροή ώστε η CIA θα πάρει την δική της πρωτογενή αλυσίδα ροής δεδομένων και ενδεχομένω και άλλα τμήματα της Αμερικανικής του Αμερικανού Συστήματος Συλλογής Πληροφοριών. Αν δούμε λοιπόν τι στοιχεία είχε ο Σνόουντεν πρόσβαση σε αυτά, ίσως δεν είχε στοιχεία α, που να αφορούν μια συγκεκριμένη αποστολή της CIA και μόνο. Αλλά αν μπορούν να παίρνουν αντίγραφα οι υπηρεσίες ασφαλείας χωρίς καμία μορφή περιορισμού γιατί έχουν ήδη φιλτραριστεί και αφορούν υποτίθεται μόνο ξένους. Το επόμενο σημείο είναι η σελίδα 23 σε σχέση με τα δικά μας εργαλεία προστασίας δεδομένων που προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι με το Safe Harbor, με τις άλλες διαδικασίες και επίσης για το θέμα του υπολογιστικού νεύους. Μια παρατήρηση που θέλω να κάνω εδώ και είναι πολύ σημαντική είναι ότι υπάρχουν παραθυράκια. Φαίνεται ότι στα τελευταία 10 χρόνια οι υπάλληλοι της Κομισιόν με τη γνώση τους ή χωρίς να το ξέρουν έχουν δεχθεί να υπάρχουν παραθυράκια που λένε εθνική ασφάλεια, αλλά αυτό σημαίνει την εθνική ασφάλεια των κρατών μελών ή την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Και επίσης υπάρχει η φράση νομικά δεσμευτική αίτηση. Για τους Αμερικανούς καλύπτει αυτό όλες τις μορφές συλλογής δεδομένων, ακόμα και συλλογή δεδομένων για πολιτικούς στόχους. Θα ήταν σημαντικό λοιπόν για την Επιτροπή σας να επανέλθει στα έγγραφα της Κομισιόν τα τελευταία δέκα χρόνια για να αναλύσει ποιος έχει κάνει αυτές, πάρει αυτές τις αποφάσεις. Έγινε καλή την πίστη, υπήρξε ασχετοσύνη, υπήρξε συνενοχή. Θα πρέπει να το ψάξουμε αυτό. Στο τέλος της σελίδας 24, τα έχω παρουσιάσει αυτά ίσως με πιο ομό τρόπο και αν προχωρήσουμε τώρα σε κάποιες από τις συστάσεις, τις προτάσεις μου. Όταν έκανα αυτές τις συστάσεις γνωρίζω ότι έχετε ζητήσει να επαναφερθεί το άρθρο 42, αλλά προτού φτάσω εκεί παρουσίασα την ιδέα ότι όπως είναι τώρα τα πράγματα και όπως τα καταλαβαίνουμε, οι πολίτες των της Ευρωπαϊκής Ένωσης θέτουν σε κίνδυνο τα στοιχεία τους χρησιμοποιώντας αμερικανικές ιστοσελίδες. Η οδηγία 9546 ζητά να υπάρχει πληροφόρηση για όλους τους κινδύνους όταν κανείς θέτει τα στοιχεία του αυτά σε μια ιστοσελίδα. Υπάρχουν λοιπόν οι εξουσίες που θα δίνουν τη δυνατότητα να πληροφορούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες ότι αν χρησιμοποιήσουν αμερικανικές ε, ιστοσελίδες, τότε θα χρησιμοποιούνται από τις Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Αν γίνει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον θα ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ποια είναι η πραγματικότητα. Και ίσως και οι Αμερικανοί θα ξανασκεφτούν, αλλά αυτό θα μπορούσε να έχει ένα πολιτικό αποτέλεσμα, θα αυξήσει τη συνειδητοποίηση και ίσως την πολιτική ε, αλληλεγγύη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εξάλλου είναι σαφές από την ανάλυση αυτή ότι οι κύριοι μηχανισμοί που έχουμε για την εξαγωγή δεδομένων δεν είναι προστατευμένοι εναντίον της νομοθεσίας Patriot ή Pfizer. Δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχει κάποιος λόγος να συνεχίσουν οι μετα... μεταφορές πληροφοριών φάση του Safe Harbor ή άλλων συστημάτων. Φυσικά πρέπει να σταματήσουμε, αν το σταματήσουμε πρέπει να το σταματήσουμε ένα στρατηγικό και βαθμιαίο τρόπο, γιατί αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Θα ήταν λοιπόν πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς μπορούμε εμείς να αναπτύξουμε μια σοβαρή βιομηχανική πολιτική για ένα ευρωπαϊκό υπολογιστικό νέφος. Και όταν φτάσουμε στην επόμενη έκθεση για τις αστηριότητε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια κρατημέλη θα βρεθούν σε προβληματική θέση. Αν δούμε λοιπόν τα θέματα του άρθρου 42, υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη στη σελίδα 28. Ο επικεφαλής της Yahoo είπε πρόσφατα ότι αν είχαν πει περισσότερο για την πίεση που υπέστησαν βάσει του 702, θα μπορούσε αυτοί και οι συνεργάτες να πάνε στη φυλακή για κατασκοπία τουλάχιστον 10 χρόνια και ενδεχομένως μέχρι 30 χρόνια ή ακόμα και θανατική ποινή. Δεν σας λέω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό, σας λέω ότι υπάρχει στην Αμερικανική νομοθεσία. Όταν υπάρχει μια τέτοια ποινικοποίηση λοιπόν, εμείς θα δημιουργήσουμε μια σύγκρουση νομική με το άρθρο 42 όταν στο, στην ευρωπαϊκή πλευρά θα πληρώνει κανείς 2% πρόστιμο ενώ από την άλλη μεριά επαπειλείται μια ποινή 30 ετών. Λοιπόν, από την εμπειρία μας με τη Microsoft, μια ένα τέτοιο πρόστιμο δεν θα κάνει τίποτα. Θα πρέπει αλλιώς να κάνουμε τη μη συμμόρφωση με το Άρθρο 42 πάρα πολύ σοβαρό ποινικό αδίκημα. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το κανονισμό, τα κράτη-μέλη έχουν απόλυτη διακριτική ευχέρεια να θέτουν πρόστιμα για αυτή την ε, παράβαση. Θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, να πούμε ότι είναι ένα σοβαρό ποινικό αδίκημα και επίσης το επίπεδο των ε, προστήμων που προτείνονται είναι πάρα πολύ ανεπαρκές. Ξέρω πολύ καλά μια περίπτωση. Η Microsoft ε, έλαβε ένα, της επευλήθη ένα πρόστιμο ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων για μια υπόθεση που έχει να κάνει με τοπικά δίκαια. Αλλά τα κέρδη που έβγαλε η Microsoft με την παραβίαση αυτή που έκανε ήταν περίπου 20 δισεκατομμύρια. Επομένως κάποιος ο οποίος κάνει ένα ψυχρό και κοινικό υπολογισμό δέχεται το πρόστιμο του ενός δισεκατομμύρια για να βγάλει τα 20 εκατομμύρια. Γι' αυτό, δισεκατομμύρια. Γι' αυτό πιστεύω ότι για να μπορούμε να έχουμε μια πραγματική στρατηγική και να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με το άρθρο 42 θα πρέπει να αυξηθούν τα πρόστιμα τουλάχιστον 10% μέχρι το 20%. Μπορεί να σας φαίνεται υπερβολικό αυτό, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτοί, αυτές οι εταιρείε έχουν τόσο μεγάλους πόρους και τόσο ισχυρές επιχειρηματικές στρατηγικές που πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, την αύξηση αυτή των προστήμων. Το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι από τότε που ξέρουμε για το σύστημα αυτό της NSA να υπονομεύσει συστήματα κρυπτογράφησης, αλλά δεν ξέρουμε πια, το άρθρο 42 θα αφορά διαδικασίες, αλλά όχι αυτούς που πουλάν συστήματα ασφαλείας. Θα πρέπει να ζητήσουμε το άρθρο 42 να αφορά και αυτούς. Αν η NSA τους υποχρέωσε να βάλουν κάποιο δούριο ύπο στα προγράμματά τους, θα πρέπει να το πούν στην Ευρωπαϊκή Ρυθμιστική Αρχή. Επομένως, δημιουργούμε άλλη μία ε, σύγκρουση ανάμεσα σε δύο νομοθετικά συστήματα και επομένως είναι σε δύσκολη θέση αυτές οι εταιρείε αν συμμορφωθούν με τον Αμερικανικό νόμο και όχι τον Ευρωπαϊκό νόμο. Θα σταματήσω εδώ για ερωτήσει και δεν ξέρω αν έχετε κάποια συγκεκριμένα θέματα που θέλετε να θίξετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τον εισηγητή μας, τον Κλοντ Μωράης. Κύριε πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω μας ξυπνήσατε όλους νομίζω με αυτή την τελευταία συνεδρία. Ήταν εξαιρετική επίδοση. Ε, ήταν πολύ σημαντική η ανάθεση αυτής της έκθεσης, ε, γιατί χρειαζόμαστε μια στρατηγική αξιολόγηση του τομέα που είναι πολύ πλοκός, ε, δεν είμαστε όλοι δήμονες σχετικά και χρειαζόταν μια στρατηγική έκθεση. Βέβαια εσείς παραδεχθήκατε ότι είναι ταχαίως μεταβαλλόμενη όλη η κατάσταση. Οπότε ακόμη και αν προβούμε σε στρατηγικές αξιολογήσεις ή συστάσεις, ενδεχομένως να μας ξεπεράσουν τα γεγονότα. Πάντως ε, αυτό πρέπει να το κάνουμε και ήταν μια έρευνα άλλωστε σύντομη χρονικά. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να έχουμε μια επισκόπηση του όλου αυτού τομέα γιατί γίνεται έρευνα. Εσείς λοιπόν πολύ ε, μέσα στην προθεσμία κάνατε ό,τι έπρεπε. Εγώ δεν διάβασα όλη την έκθεση, διάβασα κάποια κομμάτια της μπορούν οι συνάδελφοι να τη διαβάζουν σιγά σιγά και όσο ενημερωνόμαστε νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη δράση μας πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Στη σελίδα 27 ε, μας αναφέρεται ποιες είναι οι στρατηγικές μας επιλογές ως Κοινοβούλιο. Και νομίζω ότι ακριβώς αυτό θα πρέπει να είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω ούτε θέλω τίποτα, αλλά μια από τις μεγάλες συστάσεις. Εγώ βέβαια μπορώ να σας κάνω ερωτήσει για οποιοδήποτε κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, η άμεση δήλωση που κάνατε ήταν πάρα πολύ ειλικρινής, πάρα πολύ σαφής και η όλη ιδέα ότι δηλαδή και αν γίνει με τα ηλεκτρονικά μέσα Ενημέρωση θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές επιπτώσεις και για τη δημόσια ζωή, αλλά και ε, σε οποιοδήποτε ε, κομμάτι της προσωπικής ζωής ε, των ατόμων. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αλλά σε έρθω τώρα στην ουσία, στις συστάσεις που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Για το cloud computing, για παράδειγμα, υπάρχει ένα αίτημα 702 φάσα και νομίζω στην έκθεση σας λέτε ότι θα θα συμβεί, άρα θα περάσουμε στο ευρωπαϊκό cloud computing. Αυτό λέτε στην ε, έκθεσή σας ουσιαστικά. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, σας κάνω το εξής ερώτημα. Πράγματι υπάρχουν ε, πιθανότητες να έχουμε ευρωπαϊκό cloud computing. Ξέρω ότι συζητήσατε στις διάφορες ε, ανταλλαγές που είχατε και για το παράδειγμα της Βραζιλίας. Οι Βραζιλιάνοι, μίλησε και η Άννα πριν, μιλάνε για διατήρηση των δεδομένων εντός της χώρας ε, και μέσα στην επικράτειά τους. Πώς θα δουλέψει αυτό. Έρχεται σε αντίθεση με αυτό που είπατε, δηλαδή ότι αν αυτό συμβεί θα ξεπεραστεί από άλλη τεχνολογία. Θα παρακαμφθεί ή μπορεί να υπάρξει σεβασμό στην εθνική κυριαρχία. Κάποια άλλα θέματα που έχετε θέσει στις δαρτικές σας επιλογές. Κρυπτογράφηση. Είχαμε ακούσει από διάφορους τι γίνεται με την ε, κρυπτογράφηση NSA, HGQ λοιπά, Βρετανική υπηρεσία, Αμερικανική υπηρεσία. Εσείς λέτε είναι ένας τεχνολογικός τομέας. Συστάσεις μπορούμε να προβλέψουμε σε αυτή την έκθεση για να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το τεχνολογικό κλάδο. Υπάρχει κάτι χρήσιμο εδώ, για μας εδώ στο Κοινοβούλιο. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε στο Κοινοβούλιο αυτό το τεχνολογικό κλάδο και αυτό να μας βοηθήσει. Πού θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για μας αυτή η έκθεση, αφού ασχολείται και με τεχνολογία και με πολιτική. Νομίζω ότι τον Ιανουάριο 2014 θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει με την έκθεση για να έχουμε διαμορφώσει κάποια εικόνα για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε, για το ποια θα είναι η μελλοντική μας πολιτική και με τα θέματα πολιτικής και με τα θέματα της τεχνολογίας. Γιατί μπορεί κανείς να είναι παροχημένος μέσα σε εβδομάδες ή μήνες. Ο Άξελ Φως. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι έχετε πει στις, ε, γιατί αν αυτό που είπατε για τις αμερικανικές αρχές ισχύει και για τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Και θα ήθελα να έχω τη δική σας άποψη ότι αν κάνουμε συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ίσως και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάλι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε κάτι αντίστοιχο με την Κίνα ή με τη Ρωσία ή άλλα μέσα πίεσης. Έχετε κάποιες ε, <clears throat> ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και επίση αυτά που λέτε για το Safe Harbor, το σύστημα αυτό στο κείμενό σας. Τα βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που είπατε για το άρθρο 42 και τα πρόστιμα της ε, ποινές που μπορεί να επιβληθούν και για το Safe Harbor. Είναι το ερώτημα είναι γιατί έχουμε αυτή τη συμφωνία με τις ΗΠΑ, με άλλες χώρες δεν έχουμε κάποια τέτοια συμφωνία. Όλοι μας είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε το σύστημα αυτό Safe Harbor να το καταγγείλουμε ή να βρούμε άλλες συμφωνίες οι οποίες έχουν τα σωστά πρότυπα. Αλλά δεν ξέρω τι γίνεται με άλλες χώρες αν μπορούμε να έχουμε αντίστοιχες συμφωνίες. Ε, άκουσα ότι η να βρουμε αλλες συμφωνιες οι οποιες εχουν τα σωστα προτυπα αλλα δεν ξερω τι γινεται με αλλες χωρες αν μπορουμε να εχουμε αντιστοιχες συμφωνιες ακουσα οτι η κινα παράγει υπολογιστές οι οποίες έχουν ήδη κάποιο λογισμικό παρακολούθησης μέσα. Αυτά τα πράγματα είναι γνωστά, ε, πώς τα αντιμετωπίζετε. Δεν θα μιλήσω εγώ, θα μιλήσω τελευταία, ο Γιάνν Άλμπρεχτ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την γενική αυτή περιγραφή της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής μελέτης. Νομίζω ότι Έχω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για την προστασία του πληροφοριδότη που βάλατε κι εσείς ως ένα, μια σημαντική σύσταση. Με κάτι που βέβαια πρέπει να συζητήσουμε και όπου θα ήθελα να γνωρίζω ποιες θα ήταν οι πραγματικές πιθανότητες να γνωστοποιηθούν οι παραβιάσεις αυτές ή η οι ε, παράνομες συμπεριφορά και πώς μπορούμε αυτό να το περιορίσουμε στο θέμα της ασφάλειας των δεδομένων. Το δεύτερο θέμα αφορά την βιομηχανική πολιτική για το ευρωπαϊκό σύννεφο. Αν μιλάμε λοιπόν για τις δυνατότητες, πώς μπορούμε να ενεργήσουμε, υπάρχουν πολλές πολιτικές, πολλές, πολλά ερωτήματα για το τι μπορούμε να κάνουμε νομικά, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει απειλή. Υπάρχει πιθανότητα πραγματικά να φτιαχτεί ένα ευρωπαϊκό σύννεφο, νέφος. Και τέλος, το θέμα της συζήτησης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, που βεβαίως είναι και πιο σημαντική για μας εδώ. Υπάρχουν κινήσεις σε σχέση με την πολιτική συζήτηση ή αλλαγές όπου θα μπορούσαμε ήδη να εστιάσουμε και να πιέσουμε την Αμερικανική πλευρά αν υπάρχουν δηλαδή κάποιε τάσει, θα μπορούσαμε και τάσεις για αλλαγή, θα μπορούσαμε και εμεί να ασκήσουμε κάποιες πιέσει προς του εταίρου μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ. Καταρχήν με ενδιαφέρει όλη αυτή η προβληματική των μέτρων κυρώσεως των ποινών που μπορούν να επιβληθούν. Υπάρχουν κάποιες προτάσεις που ήδη συζητούνται μεταξύ μας ως κοινοβούλιο που έχουν σε στόχο μία όξυνση των ποινών, αλλά φυσικά εσείς λέτε ότι δεν επαρκεί αυτό. Πώς θα έπρεπε να αντιμετωπίσει κανείς αυτά τα πράγματα. Τα βλέπετε μόνο σε επίπεδο <clears throat> ποσοτικό ή βλέπετε και δυνατότητα να υπάρξει μια ποιοτική αλλαγή, να αντιμετωπισει κανεί αυτα τα πραγματα τα βλεπετε μονο σε επιπεδο ποσοτικο η βλεπετε και δυνατοτητα να υπαρξει μια ποιοτικη αλλαγη να εχουμε μια πιο δεσμευτική νομοθεσία για τα θέματα αυτά. Δεύτερο σημείο, λέτε ότι δεν υπάρχει καμιά αποστασία και κανένας περιορισμός παρακολούθησης για τους μη Αμερικάνους. Πού μπορεί να εδρεωθεί ένας υπερεθνικός διάλογος για τα θέματα αυτά. Είναι τόσο σημαντικό το θέμα αυτό για την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών που δεν είναι Αμερικανοί. Πώς μπορούμε λοιπόν να φανταστούμε ένα τέτοιο διάλογο και να έχουμε μια δυνατότητα να συζητήσουμε σε ένα επίπεδο ισότητας με τους Αμερικανούς. Και επίσης αυτά που είπατε για τους πληροφοριοδότες, τους whistleblowers που καταγγέλνουν κάτι. Δεν θα πρέπει να έχουμε κάτι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την προστασία αυτών των ανθρώπων. Και τέλος ένα ευρωπαϊκό σύστημα για υπολογιστικό νέφος. Μπορεί να γίνει αυτό Φυσικά αυτό είναι μια, ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε για τις εναλλακτικέ λύσεις. Ευχαριστώ. Παίρνω και εγώ τώρα το λόγο πρώτα απ' όλα για ένα ευρωπαϊκό νέφος. Φαίνεται σαν να είναι αντιφατικό αφ' αυτού το σύννεφο, το νεύος αυτό είναι μεγάλο, σε όλη τη δυναμικότητα, τη χωρητικότητα. Εγώ δεν είμαι και πολύ μεγάλος οπαδός του να περιφράξουμε την Ευρώπη, αν θέλετε, κατά κάποιο τρόπο και να μην εκμεταλλευτούμε τις νέες ε, βέβαια ε, δυνατότητες μας προσφέρει τεχνολογία, αλλά το να έχουμε ένα αντίβαρο απέναντι στην αμερικανική κυριαρχία στην αγορά δεν είναι κακή ιδέα ώστε να γίνουμε πιο σημαντικοί και πιο ισχυροί σε αυτό το νέφος μέσα, γιατί και αυτό είναι το ερώτημά μου προς εσάς. Ακόμη και αν βάλουμε ένα φράκτη γύρω από την Ευρώπη, θα έχουμε ένα 100% ευρωπαϊκό νέφος, αλλά αυτό δεν θα σημαίνει ότι αυτόματα τα δεδομένα δεν θα μπορούν ε, να τα αποκτήσουν ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι Αμερικανοί. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, είναι και νομικό το ζήτημα. Οποιαδήποτε εταιρεία, α πούμε ότι έχουμε μια εταιρεία που είναι μέσα στο ευρωπαϊκό νέφος, αλλά ε, μπορεί να έχει ένα γραφιάκι στις Ηνωμένε Πολιτείε, εκεί λοιπόν εμπίπτει στην ε, δικαιοδοσία την Αμερικανική. Και όχι μόνο το συγκεκριμένο της παράρτημα, αλλά και όλη η εταιρεία, όποια βρίσκεται. Δεν είναι μόνο δηλαδή φυσικό ε, το θέμα γεωγραφικό. Κατά την άποψή σας τώρα, θα ήταν δυνατόν ή εφικτό για την Ευρώπη, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την εφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων για να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι ναι. Η Κομισιό νομίζω ότι δεν δείχνει αρκετή τόλμη, δεν αξιοποιεί πλήρως ε, τις δυνάμεις της, τις εξουσίες που έχει, γιατί η τρέχουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επέτρεπε να γίνονται οι πρακτικές που βλέπουμε σήμερα. νέα, νομοθεσία εντάξει θα πρόσθεται περισσότερη ε, προστασία αλλά θα μπορούσε να βοηθήσει κατά την άποψη σας και ισχύουσα νομοθεσία. Τελευταία ερώτηση. Κάποιες φορέ κατηγορούν του Αμερικανούς, ε, αλλά μας λένε κάντε τα ίδια. Άρα, ρώτηση, έχουμε κι εμείς στην Ευρώπη ίδιους νόμους, παρόμοιους νόμους. Θα ξεκινήσω με το θέμα του νέφους γιατί είναι το πιο δημοφιλές. Προσπάθησα να προβλέψω όσο γινόταν πολλά από τα ερωτήματα περί νέφους στη σελίδα 32 στα σημεία 1-2-3 ε, και κατά κάποιο τρόπο θα σας τα διαβάσω γιατί πιστεύω πως ε, άμεσα αφορούν αυτά τα θέματα. Το, το κύριο γεγονός όσον αφορά τη ε, δεδομένα στον, υπολογισμό, στους υπολογιστές cloud. Στην ουσία τι κάνουν αυτοί οι υπολογιστές που είναι σε μια τεράστια αίθουσα, αποθηκεύουν στοιχεία και τα επεξεργάζονται. Μπορούν να τα επεξεργαστούν μόνο αν είναι αποκρυπτογραφημένα. Αν είναι κρυπτογραφημένα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, απλώ τα αποθηκεύεις. Ο πάροχος του σύννεφου λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζει τον ε, κωδικό για να μπορεί να κάνει υπολογισμούς ώστε να αποκρυπτογραφήσει και άρα να τα βάλει σε αυτούς τους τεράστιους υπολογιστές όπου θα τα επεξεργαστούν. Τότε είναι ευάλωτα τα στοιχεία σε διαταγή 702. Άρα η... Αλλά εδώ δεν υπάρχει λύση γιατί η κρυπτογράφηση είναι περιττή. Υπάρχουν κάποιες λύσεις που είναι 100.000 φορές πιο αργές όμως και δεν υπάρχει προοπτική στην έρευνα για κάτι άλλο. Καμία. Και μάλιστα οι εταιρείε δίχως ντροπή παραπλανούν την αγορά. Δεδομένω αυτή τη πραγματικότητα είναι να μένουν κλειστά αυτά τα στοιχεία ε, στον έφο μόνο στη δική σου δικαιοδοσία. Στη σελίδα 32, στο σημείο 3, μόνο αν μια εταιρεία θεωρητικά δεχτεί εντολή 702 θα μπορούσε να τα αποκρυπτογραφήσει. Αυτό θεωρητικά είναι πολύ δύσκολο γιατί το προσωπικό και η διεύθυνση θα προσπαθούσε να βρει διαφορετικούς τρόπους να διαμαρτυρηθεί, να καταγγείλει και να θέξει το θέμα από την ευρωπαϊκή νομική άποψη. Και έπειτα μια ευρωπαϊκή εταιρεία δεν, δεν θα κατηγορηθεί εύκολα για κατασκοπία. Από την άλλη πλευρά, αν δει κανεί πόσο εγκατεστημένη είναι στην ΣΥΠΑ μια εταιρεία, δεν θα πω ποια εταιρεία είναι, αλλά είναι εξαπλωμένη στη ΣΥΠΑ, ε, ε, λένε πως ε, στείλαν τα στοιχεία στη ΣΥΠΑ. Πρέπει να αναζητήσετε την ευρωπαϊκή εταιρεία που κάνει πολλά βήματα ώστε να απομονώσει τα στοιχεία, αλλά και νομικώ να απομονωθεί. Υπάρχει όμω μεγάλη διαφορά ανάμεσα στι δύο περιπτώσει. Ε, η το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχει τεράστια διαφορά όσον αφορά την ε, ασφάλεια έκθεσης από τεχνική άποψη, δηλαδή το να τους δίνεις έτοιμα τα στοιχεία ή το να μπορεί κανείς να ανοίξει μια βρύση οπτικής σύνα και να πάρει τα στοιχεία μαζικά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα, κινδύνου ανάμεσα σε αυτό το θέμα και άλλο είναι να έχει κανείς τα στοιχεία σε ένα ευρωπαϊκό ε, κέντρο αποθήκευσης στοιχείων και να πρέπει NSA να το διαρρήξει, να διαρρήξει διάφορα επίπεδα άμυνας και μετά να δει και πώς θα τα πάρει αυτά τα στοιχεία για να τα φέρει στην NSA. Στο ένα είναι πρέπει, το δίνεις έτοιμα στο πιάτο ας πούμε τα στοιχεία, ενώ η άλλη περίπτωση δυσκολεύει. Βέβαια, αν αναλύσουμε τις καταστάσεις, το πρόγραμμα της ε, Κομισιόν ήταν να φτιάξει κάτι αντίστοιχο με τον έφος, να μπορεί να εξάγει τα στοιχεία, να τα δώσει έτοιμα στο πιάτο τους Αμερικανούς και, να τα, και το άλλο, η άλλη επιλογή θα ήταν να διατηρηθούν εντός της Ευρώπης όπου θα ε, προστατεύονταν από επιθέσεις. Σύμφωνα όμως με τον νέο κανονισμό και τη διατύπωση, αυτές οι καταστάσεις ε, περιγράφονται ότι, ότι αντιστοιχούν και είναι προφανές για τον κοινό νου και για πόσο μάλλον για έναν ειδικό ε, των υπολογιστών ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι λάθος ο κανονισμός όπως έχει διατυπηθεί. Τελείως πρέπει να ξαναδιατυπωθεί κυρίως όσον αφορά τους κανόνες για την επεξεργασία των στοιχείων. Γιατί διαφορετικά θα γίνουμε ακόμα πιο ευάλωτοι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο. Να στραφώ σε κάποια άλλα ερωτήματα. Uh, if I start uh, with Mr. Να επανέλθω με την ερώτηση του κυρίου Βόσ για την κατάσταση με τη ΣΥΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν κατάλαβα ακριβώ τι εννοούσατε. Πάντως σίγουρα εγώ δεν είχα προσωπική πείρα από τη Ρωσία ή την Κίνα σε αυτό το τομέα. Νομίζω πως ούτε καν έχω δει την, γερμανική, την κινέζικη νομοθεσία. Οι Ρώσοι υπέγραψαν τη σχετική νομοθεσία, αλλά δεν θα το σχολιάσω άλλο. Τώρα για τον ασφαλή λιμένα θα πρέπει να δούμε τον, το ότι η ε, ασφαλής λιμένα στην ουσία έχει σπάσει. Χθες παρακολούθησα μία σχετική συνεδρίαση μαζί με τον κύριο Νέμις και τον ρώτησα αν θα ήθελε αυτή η συζήτηση να μείνει απόρριτη. Μου είπε όχι. Οπότε να σας πω ποια ήταν η εντύπωσή μου από αυτή την συνεδρίαση εκείνης της ομάδας όπου συζητούσαν και λέγανε ότι πρόκειται για μια εμπορική συμφωνία και δεν βλέπουν καμία, κανένα περιορισμό για πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Έτσι το βλέπουν αυτή την συμφωνία. Και πρέπει να ρωτήσουμε πώς γίνεται πριν από 13 χρόνια στην Ευρώπη να κάνουμε ένα τέτοιο τεράστιο λάθος, να είμαστε τόσο δηλαδή παραπλανημένοι, αποπλανημένοι. Τι πήγε λάθος. Δεν πρέπει να το ξέρουμε για να μην ξανακάνουμε το ίδιο λάθος το ασφαλές, ασφαλής λιμένας δεν, έχει, δεν, δεν ισχύει πλέον και σίγουρα δεν μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για οτιδήποτε κάνουμε στο μέλλον. Για να επανέλθω τώρα στην ερώτηση της κυρίας Μωράης, ε, του κυρίου Μωράης, με συγχωρείτε. Για αυτή τη φράση που κυκλοφορεί ιδιαίτερα για τη Βραζιλία, της βαλκανοποίησης, βαλκανοποίησης Του ίντερνετ. Ε, προέκυψε και στις παρατηρήσεις ε, του κυρίου Κάμερον Κέρι του Υπουργείου Εμπορίου πριν από κάνα μήνα. Νομίζω ανοησίες είναι αυτά. Εδώ δεν μιλάμε για ε, λογοκρισία, λέμε για περιορισμένη πρόσβαση στα στοιχεία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Όχι, μιλάμε για διευκολύνσεις και υπηρεσίες και εταιρείε τοπικά στην Ευρώπη και να καλέσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες να χρησιμοποιούν. Δεν υπάρχει υποχρέωση, είναι επιλογή. Αν κάποιο θέλει να στείλει τα στοιχεία του που υπάρχουν στα χέρια της NSA, κανένας δεν λέει να το σταματήσει αυτό, με, άμα κανείς ε, δώσει τη συγκατάθεσή του, και το αποφασίσει ο ίδιο, Ωστόσο, θα έπρεπε να μην είναι δυνατόν, είτε πρόκειται για κυβερνητική οργάνωση, είτε για ιδιωτική οργάνωση, από τη στιγμή που θα έχουν πάρει τα δικά σου στοιχεία, να αποφασίζουν μετά πού θα τα στείλουν ή αν θα τα στείλουν κάπου αλλού. Αυτό θα πρέπει να πάψει, να σταματήσει με μια πολύ πιο ξεκάθαρη διαδικασία έγκρισης, αδειοδότησης. Και αυτή η ιδέα της βαλκανοποίησης δεν νομίζω είναι ανοησία. Μιλάμε για αύξηση των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων ώστε τα άτομα να μπορούν να προβαίνουν σε επιλογές όντας ενημερωμένα. Το θέμα τώρα της ε, κρυπτογράφησης είναι πολύ σοβαρό διότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε την ε, κρυπτογράφηση χρησιμοποιούσαμε μέχρι πριν τρεις μήνες, πριν τις αποκαλύψεις δηλαδή, οι επικεφαλής της ασφάλειας εξακολουθούν να ε, πιστεύουν ότι η βασική τεχνική, ο βασικός αλγόριθμος εξακολουθεί να λειτουργεί. Όμως πριν από τρεις εβδομάδες ο βασικός ε, πολιτής ε, λύσεων ασφάλειας στον κόσμο, τα εργαστήρια RSA, είπαν ότι το βασικό τους προϊόν για εντοπισμό βασιζόταν σε έναν ε, σε ένα νούμερο, σε ένα στοιχείο που έλεγε, το οποίο μάλλον είχαν ε, βρει η NSA. Το έλυσε η NSA. Άρα οι ίδιοι είπαν μην αγοράζετε το προϊόν μας, μην το χρησιμοποιείτε το προϊόν μας, γιατί δεν είναι πια ασφαλές. Ε, το θέμα της ασφάλειας είναι δύσκολο, τόσο για το software όσο και για το hardware. Το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο για τους ε, πολιτές, ε, τους ε, φορείς στο mainstream, τους μεγαλύτερους δηλαδή. Έχουν κάποια σχέση με την Εθνική Υπηρεσία Ασφάλειας των Αμερικανών. Πάντως πιστεύω πως θα έπρεπε να ευνοούνται πάντοτε οι λύσεις, οι ανοιχτές, δωρεάν. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε την αρχιτεκτονική ασφαλείας, αλλά θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί όσον αφορά τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε. Νομίζω πως απάντησα. Παρακαλώ, αν κάτι ξέχασα, να μου το θυμίσετε. Ωραία. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στο δεύτερο γύρο. Έχω τρεις συναντές που έχουν στήσει το λόγο. Ρομέρο, Βάινχολτσερ, Μορβάη. Κάποιος άλλος. Then it will be those three. Κύριε, Ρομέρο, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον ε, κύριο Μπάουντεν. Ε, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Αν θυμάστε καλά, σας είχαμε δει όταν παρουσιάσαμε τις τροπολογίες μας για την νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Και είχαμε συμπεριλάβει μια τροπολογία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε ορισμένα από τα προβλήματα με το νέφος αυτό. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, της υποχρεώσεις ε, των υπεργολάβων οι προμηθευτές έχουν τις επιχειρήσεις τους οποίους, τις επιχειρήσεις οποίες ε, προσλαμβάνουν και που ε, λέμε ότι είναι ένα νέφος για να μην ξέρουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ξέρουμε όμως ότι είναι υπεργολάβοι εταιρείε αυτών των μητρικών εταιριών. Έχουν υποχρέωση να τηρήσουν ε, τις ίδιες ή μάλλον αν έχουν την υποχρέωση να τηρούν ακριβώς ε, τις ίδιες ε, απαιτήσει ε, και να πληρούν τις ίδιες προποθέσει, μήπως αυτό είναι μια λύση. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να είναι μια απάντηση και αν ναι, πόσο επαρκή θα μπορούσε να είναι. Γιατί και στην Ευρώπη θα μπορούσαν να υπάρχουν πολλέ εταιρείε νέφη κατά κάποιο τρόπο που όμω θα ήταν υποχρεωμένε να εφαρμόσουν την ίδια νομοθεσία. Έχουμε το άρθρο 42 της ρήτρα κατά της ε, φύσα, αντιφύσα. Ακούσαμε κάποιες ε, ειδήσει ότι αφορά τις ε, εξουσίες των επιχειρήσεων και ανασχολή της κυρίας Ρέντινγκ πυρητή συγκατάθεση, συνένωση που είναι ένα πολύ σημαντικό. Αν έχουμε σε αυτό τον άξονα της προσέγγισης δεδομένων δυσκολίες, όπως ένα άξονα είναι αυτή η ρητή συνένεση, τότε σε αυτό το άρθρο 42 θα έχουμε επίσης δυσκολίες. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, αρκεί όπω έχει διατύπωση το άρθρο 42 σήμερα, αν δεν διαγραφεί, για να γίνει αυτό που εσεί μας προτείνετε, δηλαδή δεν θα μπορούσαν να μεταφέρουν σε τρίτες χώρες αν δεν υπάρχει ε, η πρώτερη συνένεση της εταιρείας ε, δεν θα μπορούσαν να διαβάσουν δηλαδή τότε τα, τα στοιχεία. Και αν ναι, αν ισχύει αυτό, εμείς δεν έχουμε μια ε, αρχή εποπτείας δεδομένων, γιατί το Συμβούλιο το οποίο δημιουργείται δυνάμει αυτού του νόμου για την προστασία δεδομένων δεν έχει αρμοδιότητες. Ίσως όμως θα μπορούσε κάποιο κράτος μέλος που έχει αρμοδιότητες ε, να θέσει ένα τέτοιο ζήτημα. Δεν ξέρω, είναι δυνατό αυτό. Γιατί αν όχι, πρόεδρος μπορείτε να ολοκληρώσετε. Κύριε Ρωμέ, αν μπορείτε, ε, απαντήστε μου. Ναι. Συγγνώμη, αλλά ήθελα να έχω μια απάντηση σε ό,τι αφορά αυτή τη ρήτρα αντιφύσα. Αν δεν αλλάξουν τους νόμους τους οι Αμερικανοί θα είναι δύσκολο. Ναι, για να ακούσουμε και άλλους, ε, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα. <clears throat> Έχουμε αρχίσει να παρακολουθούμε πως ε, η διατλαντική ομάδα έχει μια εποπτεία της κατάστασης και θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι τα έγγραφα τα οποία δίδονται σε αυτές τις διατλαντικές ομάδες. Η δική μου εντύπωση είναι ότι υπάρχει πάλι ένα ψηφιακό χάσμα μεταξύ των Αμερικανών και του υπόλοιπου κόσμου. Και το ερώτημα μου είναι, πιστεύετε εμείς με το πακέτο το οποίο έχουμε εμείς μπορούμε για τα υποστασία δεδομένων μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα το οποίο μέχρι στιγμής δεν του έχουμε δώσει την πρέπουσα σημασία. Κυρία Μορβάη, τελευταίο ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ε, που ήρθατε. Ε, ποια είναι η κατάσταση σε ένα κατωμέλος το οποίο πριν να κάνει εκλογές μπορεί να καλέσει ανθρώπου που έχουν φτιάξει το λογισμικό τοπικά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αποκλειστικά το λογισμικό που έχει προετοιμαστεί από αυτούς ή μπορεί ενδεχομένω να αγοράσει λογισμικό σε μεγάλες ποσότητες και πολύ ακριβό από την Microsoft. Υπάρχουν κρατημέλη που κατέφυγαν στη χρήση λογισμικών της Microsoft έχουν προβεί δηλαδή σε στρατηγική ε, συμφωνία για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την Microsoft στη δικαιοσύνη, στην παιδεία κτλ. Κατά τη γνώμη σας, αυτό ε, περιέχει κινδύνους. Δεδομένης της σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην Microsoft και την Εθνική Ασφάλεια των ΗΠΑ, στην ουσία αυτό το κράτος δίνει τα στοιχεία του στις υπηρεσίες ασφαλείας της Αμερικής ή και σε άλλους δεδομένου ότι περνάνε όλα από τη Microsoft. Και η Microsoft είναι σε μια ιδιαίτερη θέση. Με ενδιαφέρει πολύ η γνώμη σας. Και σας παρακαλώ να μην, να μην ε, παρακάμψετε την ερώτησή μου. Κοιτάξτε. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 9546, αν σκεφτεί κανεί τον ασφαλή λιμόνα, το άτομο, μάλλον οι μεμονωμένε ε, ε, αρχές ασφαλεία δεδομένων έχουν ήδη, με βάση τα όσα έχουν δημοσιευθεί, να, ε, το δικαίωμα να σταματήσουν οποιαδήποτε ροή δεδομένων προς οποιαδήποτε εταιρεία ασφαλή λιμένα. Ωστόσο και η εταιρεία μπορεί, και κάποια συγκεκριμένη κυβέρνηση μπορεί να κλείσει μια τέτοια εταιρεία αν το επιθυμεί. Μπορεί αύριο να πάει και να το κάνει και πιστεύω πως θα πρέπει να το κάνει κιόλας. Παρομοίως, τα, οι συμβάσεις πρότυπα που έχουν συνταχθεί από την Κομισιόν από το 2001 έχουν, προβλέπουν τη δυνατότητα να άρουν και να αναστείλουν συμφωνίες γιατί η έκθεση αποδεικνύει γιατί στην ουσία επιτρέπουν την παράνομη παρακολούθηση στοιχείων από μια υπηρεσία ασφαλεία ε, άλλη χώρα. Δεν υπάρχει πλέον αμφιβολία γι' αυτό. Και γι' αυτό και δίνεται τέτοια έμφαση στο άρθρο 42, στη συγκατάθεση, στη συνένεση. Γιατί αν δεν έχουμε οποιαδήποτε άλλη διαρθρωτική συμφωνία με τη ΣΥΠΑ, τότε μόνο η συνένεση μα μένει. Εγώ αυτό που προτείνω είναι ένα είδο διπλή στρατηγική. Ε, από τη μια πλευρά δηλαδή θα αυξήσουμε την πολιτική συνειδητοποίηση και θα μειώσουμε την ε, έκθεση εκτός όταν υπάρχει πλήρως ενήμερη συγκατάθεση και από την άλλη πλευρά δημιουργούμε τις δυνατότητες για ένα ευρωπαϊκό νέφος ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε την αμερικανική ε, πολιτική και εμπορική γνώμη. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να δούμε οργανώσεις πολιτικών ελευθεριών και εμπορικά σώματα, αντί να πιέζουν για να μειωθεί η ευρωπαϊκή ιδιωτικότητα, να πιέζουν την αμερικανική κυβέρνηση για καλύτερη προστασία ιδιωτικής ζωής για τους μη Αμερικανούς. Αυτή είναι η βασική στρατηγική ιδέα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ρεαλιστές όταν πιστεύουμε, εάν πιστεύουμε πως η αμερικανική δημόσια συζήτηση ε, ε, ασχολείται με τη γνώμη μας. Εγώ έχω μετρήσει τις αναφορές και έχω παρακολουθήσει την Αμερικανική συζήτηση για το θέμα τα τελευταία δέκα χρόνια μέχρι πριν τρει μήνε και δεν ε, σα κοροϊδεύω. Μία αναφορά έχει γίνει σε δέκα χρόνια συζήτηση για το ενδιαφέρον για τους μη Αμερικανούς. Μια ψηλό αναφορά σε μια συνεδρίαση επιτροπής. Στους τελευταίους τρεις μήνες τρεις αναφορές Human Rights Watch, ο κύριος Μάρξ από το Συμβούλιο Αποπτίας ε, και ένας άλλος ε, δικηγόρος περί, ε, που ασχολείται με πολιτικές ελευθερίες. Τίποτα στο Κογκρέσο. Έχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά αν θέλουμε να παρουσιάσουμε τις ευρωπαϊκές μας απόψεις, να τις περάσουμε στη ΣΥΠΑ, να έχουμε βουλευτές, αντιπροσωπείες, υπαλλήλους που θα εμφανίζονται στα στούντιο, τα τηλεοπτικά, στην συζήτηση στην Αμερική για το θέμα αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε επαρχιώτες. Τα θέματα υπεργολαβίας. Πολύ σημαντικά. Αν τα δείτε από την άποψη ενός δικηγόρου σε μια διαδικασία ε, ε, επεξεργασίας νέφους για μια εταιρεία, που δηλαδή θα πάνε και θα αποθηκευθούν τα στοιχεία, είναι πολύ δύσκολο και η Κομισιόν προσπαθεί να τυποποιήσει συμβάσεις. Δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της συνολικής λύσης και είναι ένας μεγάλος τομέας αβεβαιότητας. Είναι το 10% της λύσης που χρειαζόμαστε αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Um, well, we talk, I've mentioned already that data protection authorities have, in my view, uh, considered. Οι ε, υπηρεσίες, οι αρχές προστασίας των δεδομένων έχουν δυνατότητες, έχουν αρμοδιότητες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή αρχές των ε, οι Ευρωπαϊκές Αρχές Εποπτείας των Δεδομένων και ο Ευρωπαϊκός Επόπτης, ο Ευρωπαίος Επόπτης, δεν έχουν κάνει τίποτα για την ώρα. Ούτε για τους ασφαλείς λιμένες, ούτε βέβαια κατά συνέπεια τα τελευταία δύο χρόνια. Τους έχει πάρει ο ύπνος στο τιμόνι και πρέπει κάποιος να τους ξυπνήσει. Και θα ήταν χρήσιμο για την Επιτροπή να καλέσει του εκπροσώπου αυτών των αρχών να μα δώσουν λογαριασμό για το τι ακριβώ κάνουν για αυτά τα θέματα τα τελευταία δύο χρόνια και να αιτιολογήσουν την αδράνειά του. Γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Ενώ είχαν τη δυνατότητα, είχαν εξουσίες για να δράσουν. Και πάλι στι συστάσει μου δεν ανέφερα συγκεκριμένε ιδέε για μεταρρύθμιση όσον αφορά τις ρυθμίσεις περί προστασίας, αρχών προστασίας των δεδομένων. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει ένας επίτροπος των λαών για να αντιπροσωπεύει με ατομικά δικαιώματα. Και, και απομακρυνόμενος λίγο από την ερώτηση που μου θέσατε, υπάρχει μεγάλη αναποτελεσματικότητα στην τεχνική ανικανότητα των αρχών ε, προστασίας των δεδομένων. Όπως γνωρίζω, μόνο καμιά δεκαριά από όλους αυτούς τους υπαλλήλους αυτών των υπηρεσιών έχουν τη τεχνική γνώση για να, να, να κάνουν προστασία δεδομένων και μόνο ένας από ό,τι ξέρω έχει πτυχίο για, ως μηχανικός υπολογιστών ειδικευμένος στην ασφάλεια και στην ιδιωτικότητα. Το 99% είναι υπάλληλοι. Φανταστείτε ένα αεροδρόμιο, α πούμε, που αντί να έχει διχμηχανικούς, ε, να έχει υπαλλήλου μόνο. Να έχουμε ποσοστώσεις. Εγώ είναι ε, κάπως ε, ψυχρό το θέμα, αλλά δεν βλέπω άλλο τρόπο να το κάνω. 25% τουλάχιστον άνθρωποι με συγκεκριμένη σταδιοδρομία για ανώτατες θέσεις είναι τόσο πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι τόσο χάλια η κατάσταση και πρέπει να δείτε το, τα περασμένα δύο χρόνια δράνειας για να καταλάβετε πόσο χάλια είναι. Oh, um, the report, Τώρα, η ομάδα εμπειρογνωμόνων τη περιβαλλοντικής ε, συνεργασία μα δεν ξέρουμε καν ποιοι είναι. Δεν έχουμε ονόματα. Αλλά ίσω γι' αυτό θα πρέπει να εκφράσουμε γενικότερα την ε, λύπη μα γιατί σε καμιά ομάδα εμπειρογνωμόνων δεν ξέρουμε ποιοι είναι, ούτε το ε, ιστορικό τους, την εμπειρογνωμοσύνη τους. Ίσως θα ήταν καλό να τα γνωρίζουμε αυτά για το μέλλον. Σε σχέση με το ρόλο της Microsoft ε, ε, στην βιομηχανία νέφους και το κλείδωμα στοιχείων, το αυτόματο, είναι αλήθεια ότι πίσω το 2008-2009 Κατά κάποιο τρόπο η βιασύνη της Microsoft που εγώ δούλευα τότε και, και είδα πραγματικά πόσο κοντά ήταν έτσι, ε, στο να το φτιάξουν. Ο λόγος λοιπόν που τόνισε τόσο πολύ το νέφος η Microsoft ήταν ότι ήθελε να προλάβει τον ανταγωνισμό γιατί αν, οι, οι πελάτες τους πήγαιναν στο δικό τους νέφος θα μπορούσαν να διατηρήσουν τη δικό τους ε, τρόπο αδειοδότησης, ε, κλειδώματο και θα συνέχισαν δηλαδή το το business αυτό ε, δεν υπάρχει υπεράσπιση γι' αυτό. Θα πρέπει να έχουν πολύ πιο στεναρή πολιτική ώστε να πάψουν αυτή το, το κλείδωμα το αυτόματο και υπάρχει μεγάλη ε, αγαθοσύνη και έλλειψη γνώσεων από πλευρά των αρχών παρακολούθησης για να εμποδιστούν αυτά τα στρατηγικά παιχνίδια που χρησιμοποιούνται κατά του κλειδώματο. Κάτι ακόμα είναι οι πληροφοριοδότες, πράγμα το οποίο δεν ανέφερα στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων. Κάποιοι θα θυμούνται ότι το Φεβρουάριο, αφού έκανα μια παρουσίαση, μου ζητήθηκε να προβώ σε κάποιες συστάσεις, ιδιαίτερα για του πληροφοριδότε, και έχουν υπάρξει κάποιε τροπολογίε που έχουν ήδη κατατεθεί, που φαντάζομαι θα τι εξετάσετε κι εσεί τον Οκτώβριο. Αυτέ οι τροπολογίε είναι εντάξει. Ε, μάλιστα πρότεινα ένα στεναρότερο πακέτο τότε το Φεβρουάριο. Υπάρχει όμω μια επιπλοκή, γιατί είναι αρκετά δύσκολο να εγγυηθούμε το άσυλο και την ε, νομική ε, για κάποιον και θα ήταν ιδανικό να μπορέσουμε να βάλουμε στον κανονισμό συγκεκριμένη ε, προστασία για τους πληροφοριοδότες. Θα βοηθούσε αυτό εδώ και σίγουρα θα χρειαστεί πολλή προσπάθεια και νομική μελέτη ώστε να διασφαλιστούν οι πληροφοριδότες. Γιατί το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στους πληροφοριδότες και θα είναι αυτοί όλοι τόσο αλτρουιστές όπως ο Έντουαρντ Σνόντεν. Μπορεί να τους ε, δοθεί κίνητρο και να, τους, ε, να θέλουν μια ανταμοιβή. Γιατί στη ΣΥΠΑ, ας πούμε, διώκονται για το υπόλοιπο της ζωής τους. Μπορεί να τους μεταγάγουν, να τους απαγάγουν και να αναγκαστούν να τρέχουν από αεροδρόμιο σε αεροδρόμιο. Με πάση περιπτώσει να έχουν μια ανταμοιβή που να μπορούν να ζήσουν κάπως φυσιολογικά τη ζωή τους αφού θα έχουν πάρει αυτή την απόφαση να δώσουν τις πληροφορίες. Αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε μια σοβαρή αποτροπή Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να Θέλετε να επανέλθετε, ναι, συγγνώμη. Δεν ξέρω αν ήταν θέμα μετάφρασης, αλλά ίσως δεν καταλάβατε καλά το ερώτημά μου. Να το ξαναπώ στα αγγλικά. Το ερώτημά μου ήταν αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος ότι αν η Microsoft αν χρησιμοποιήσουν μάλλον κυβερνήσεις το λογισμικό της Microsoft στη δημόσια διοίκησή τους κτλ. μπορεί η NSA να παρακολουθεί τι γίνεται στις ε, κυβερνητικές υπηρεσίες μέσα από το σύστημα αυτό της Microsoft και τις, τους δούριους ύπους που περιέχει. Σημαίνει αυτό ότι μια κυβέρνηση που χρησιμοποιεί ε, λογισμικό της software γίνεται τρωτή. Νομίζω ότι είναι σαφές τώρα, κύριε Μπάουντον. Είναι πιο πολύπλοκα τα πράγματα. Θα σας πω τη σύντομη Απάντηση, εγώ δεν <clears throat> εμπιστεύομαι το λογισμικό της ε, Microsoft μετά από 15 εδώ και 15 χρόνια έχω φύγει από τη Microsoft τελείως δεν χρησιμοποιώ καθόλου για τις κυβερνήσεις είναι πιο μεγάλη ανησυχία αλλά είναι μακρά η εξήγηση γιατί πολλές φορές αυτά που θεωρούν δούριους ύπους δεν είναι δούριοι ύποι υπάρχουν πραγματικοί μηχανισμοί οι οποίοι είναι πολύ πιο ε, και χρειάζεται πολύ, πολύ ώρα για να σας τα εξήγησω. Ερχόμαστε λοιπόν στο τέλος και αυτού του τμήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα στοιχεία που μας δώσατε. Το τελευταίο τμήμα της συζήτησης τώρα είναι τα συμπεράσματα του εισηγητή. Όχι, δεν θέλει να πει τίποτα ο εισηγητής. Νομίζω ότι και οι βουλευτές και όλοι μπορούν να διαβάσουν ε, τις καταλικές μου παρατηρήσεις. Um, just a couple of things, Chair. Αλλά μπορώ να σας πω και δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Κάσπαρ Μπάουντεν και τον κύριο Τσέπεσιν και τους συναδέλφους της τελευταίας συνεδρίας. Τέτοιου είδους συνεδρίες νομίζω ότι καλό θα ήταν να ακούγονταν και από περισσότερους, άξιζαν ενός μεγαλύτερου ακροατηρίου και σίγουρα θα εμπλουτίσουν πάρα πολύ και τη δική μου έκθεση αυτά που ακούσαμε. Να πω τίποτα, τη δύο λόγια για την πρωινή συνεδρία. Τι έγινε σήμερα το πρωί, αγαπητοί συνάδελφοι. Ήταν κάποια ζητήματα αυτοκριτικής ουσιαστικά. Ε, δεν πήραμε απαντήσεις για το SWIFT. Σε σχέση με αυτή την απάντηση, την επιστολή που έστειλε ο Υπουργός, ε, ο Αμερικανός, Άρα θα πρέπει να προγραμματίσουμε μια άλλη ανταλλαγή απόψεων. Επίσης υπήρχαν ε, θέματα και με την ανταλλαγή ε, με την ε, Europol και αυτό θα πρέπει να το συνεχίσουμε. Θα τα γράψω και στην εκθεσή μου. Τρίτο, το θέμα της συνεδρίασης GCHQ Belgacom τον Οκτώβριο. Πολιτικά συμπεράσματα ε, δεν θα κάνω τώρα στις καταληκτικές μου παρατηρήσεις γιατί έχουμε την έρευνα. Αυτά ήταν τα τρία που ήθελα να πω. Νομίζω, ή μάλλον όχι, δεν θα πω τίποτε άλλο. Γιατί αν συνεχίσω θα κουράσω ε, τον κόσμο και θα θέλω να φύγουν όλοι. Απλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ε, μακρά συνεδρία και να ευχαριστήσω όσους άντεξαν μέχρι το τέλος. Ο κύριος Μπρόνς νομίζω μου κάνει μια ερώτηση για την 3η Οκτωβρίου. Η συνέντευξη της 3ης Οκτωβρίου θα έχει να κάνει με την Belgacom και τους ισχυρισμούς για διεστήσεις από την GCHQ, τη Βρετανική Υπηρεσία. Θα καλέσουμε τον επόπτη, το Βέλγο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, 3 Οκτωβρίου. Το ζήτησαν οι Σκιώδης και άλλοι συνάδελφοι. Πρόεδρος, κυρία Μορβάη, θέλει το λόγο γιατί, για τη διαδικασία, για διαδικαστικό, γιατί θέλαμε να λήξουμε τη συνέντευξη. Ναι, διαδικαστικό μάλλον δύο. Στις 30, τι θα γίνει, διερευνητική συνάντηση και η αδέσμευτη μπορούν να παραστούν, ε, να είναι μέλη να την που πηγαίνει στην Ουάσιγκτον. Εγώ δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, είμαι εγγεγραμμένη. Μπορώ να πάω γιατί συζητάμε για την ε, διαφάνεια, γι' αυτό και το θέτω το ερώτημα. Πρόεδρος, ναι θα το ανακοίνω. Στις 30 του μήνα, τη Δευτέρα, 3 με 6.30, πράγματι υπάρχει μια συνεδρίαση. Θα έχουμε πρώτον μια ανταλλαγή απόψεων με την κοινότητα των πολιτών, την Αμερικανική ΕΠΗ και η Και η δεύτερη συνεδρία θα έχει να κάνει με τους whistleblowers και την νομική τους προστασία 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, αυτό που είπατε το αποφασίζουν οι συντονιστές επιτροπής. Δεν είναι νομίζω κάτι το οποίο μπορούμε να αποφασίσουμε εδώ και τώρα. Το συζητούν οι συντονιστές και φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι γίνεται πολύ λόγος, πολύ συζήτηση για την σύνθεση της συγκεκριμένης αυτής αντιπροσωπείας. Δεν είναι το δικό σας το μόνο έτοιμο. πάντως είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Just, I was just mentioning to... Έλεγα στην Πρόεδρο ότι το σχέδιο ε, καταλόγου των ακροάσεων είναι στο φακελό σας και μπορείτε να ε, προγραμματίσετε τις κινήσεις σας. Βέβαια μπορεί να αλλάξει με βάση τα αιτήματα των σκιωδών και των άλλων βουλευτών για το θέμα του SWIFT παραδείγματο χάρη που επανέρχεται από καιρού καιρό. Πρόεδρος, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλα φλέγοντα, όχι, τότε να ευχαριστήσω... Α, ο Γιάννη έχει ένα φλέγον ε, ερώτημα, πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Σε σχέση με την υπόθεση Μπελγκακόμ έχω ένα ερώτημα. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι της Βρετανικής κυβέρνησης. Απάντηση. Το έλεγξα, ναι. Η γραμματεία του Άντελος πάντων έστειλε και πάλι μια υπενθύμηση για τους Βρετανούς εκπροσώπους. Θα ενημερώσω τους Σκιώδης ευθύ αμέσω αν έχουμε πρόοδο. Αν υπήρξε σήμερα κάποια εξέλιξη. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Καλό απόγευμα.